because we are at the beginning running out of time. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. It's just uh, five. Uh, dear colleagues, dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αρχίζουμε την συνεδρίασή μας. Καλωσορίζοντας πρώτα απ' όλα την οριστήσα επίτροπο, την κυρία Γκάμπριελ, η οποία ήταν ευρωβουλευτής τα τελευταία 8 χρόνια, όπως όλοι γνωρίζετε πολύ καλά. 16 Μαΐου του 2017 ο πρόεδρος Γιούνκερ ενημέρωσε όλους εμάς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον ορισμό της κυρίας Μαρία Γκάμπριελ ως ε, επίτροπο οριστήσα με αρμοδιότητες το χαρτοφυλάκιο της ψηφιακής οικονομίας και ε, κοινωνίας. Έχουμε από κοινού αρμοδιότητα για αυτό το θέμα με την Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης. Γι' αυτό και καλωσορίζω εδώ την κυρία Κάμερβελτ. Θα συμπροεδρεύσουμε σε αυτήν ε, την σημερινή συνάντηση. Οπότε εγώ καλωσορίζω εδώ τα μέλη και των δύο επιτροπών, γιατί είναι όλοι εδώ παρόντες. Η ακρόαση αυτή θα γίνει σε ισοτιμία ανάμεσα στις δύο αυτές επιτροπές. Για να εξετάσουμε το χαρτοφυλάκιο ακριβώς της ε, οριστής σας επιτρόπου, της κυρίας Γκάμπριελ, μαζί με εκπροσώπους και της ΣΥΜΚΟ και της Γιούρι και της ΛΥΜΠΕ, των τριών αυτών κοινοβουλευτικών επιτροπών, που επίσης συμμετέχουν στην ακρόαση αυτή. Καλώς ήρθατε και εσείς λοιπόν, τα μέλη αυτών των ε, τριών επιτροπών που συμμετέχουν στην ακρόαση αυτή. Έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Σύμφωνα με τις κατευθυντήρες γραμμές που έχουμε από την ε, Επιτροπή, ο κάθε οριστής ε, επίτροπος καλείται να παρουσιαστεί για ακρόαση μπροστά στις επιτροπές εκείνες των οποίων τις αρμοδιότητες έχει και αυτός ή αυτή. Επίσης, γραπτά απαντούν σε ερωτήσεις που τους έχουν υποβληθεί προηγουμένως. Και εσείς τις έχετε τις απαντήσεις αυτές. Κυρίε και κύριοι, σας παρακαλώ, σταματήστε τις μεταξύ σας συζητήσεις. Παρακαλώ. Έχετε λοιπόν, όπως έλεγα, τις απαντήσεις της οριστής σας επιτρόπου στους φακέλους σας μαζί με την ε, επιστολή της κυρίας Γκάμπριελ, το βιογραφικό της σημείωμα και την δήλωση οικονομικών της συμφερόντων, όπως επίσης και την επιστολή της Επιτροπής Γιούρι, που ήλεγξε τα οικονομικά συμφέροντα της οριστής σας επιτροπού. Όλα αυτά τα έχετε στους φακέλους σας λοιπόν. Τώρα, επί της διαδικασίας, πολύ σημαντικό. Πρώτα έχουμε μια αρχική παρουσίαση από την οριστή οριστήσα επίτροπο για 15 λεπτά. Στη συνέχεια θα έχει και 5 λεπτά στο τέλος της ακρόασης αυτής για καταληκτικές παρατηρήσεις. Μετά τις εισαγωγικές ε, παρατηρήσεις στην αρχική παρουσίαση της οριστής σας επιτρόπου θα έχουμε χρόνο για 25 ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτές που θα γίνουν σε δύο κομμάτια. Έχουν χωριστεί σε δύο κομμάτια δηλαδή οι ερωτήσεις αυτές. Η συζήτηση θα γίνει σύμφωνα με την αρχή, τη λεγόμενη του ping-pong. Δεν ξέρω αν είναι σωστή ονομασία αυτή, εν πάση περιπτώσει έτσι το λέμε. Με πέντε λεπτά ο καθένας. δηλαδή 25 ερωτήσεις από πέντε λεπτά η καθεμία. Και κάθε φορά να το ξέρετε ότι έχουμε ένα λεπτό για την ερώτηση, δύο λεπτά για την απάντηση και υπάρχει δυνατότητα για μια δεύτερη ερώτηση από τον ίδιο αμέσως μετά με δυνατότητα απάντησης. Ένα λεπτό αυτό όμως, ε, η ερώτηση και άλλο είναι η απάντηση στη δευτερολογία. Πολύ σημαντικό λοιπόν. Ένα λεπτό ερώτηση, δύο λεπτά απάντηση και μετά ενδεχομένως, αν το αποφασίσει ο Ευρωβουλευτή, μπορεί να συνεχίσει με ένα λεπτό ερώτηση και ένα λεπτό απάντηση από την οριστή Επίτροπο. Τώρα, εκ μέρους και των δυο μας, θέλω να σας πω ότι θα φροντίσουμε να τηρείται ο χρόνος και των ερωτήσεων και των απαντήσεων. Θα είμαστε πολύ αυστηροί. Γιατί σε τρεις ώρες πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει. Η σειρά είναι ίδια με αυτήν που ακολουθούμε και στην Ολομέλεια. Η ίδια αρχή δηλαδή ισχύει. Υπάρχει διερμηνία σε 23 γλώσσες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λοιπόν τη δική σας μητρική γλώσσα Και ακριβώς θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι ό,τι θα πείτε θα περάσει από τη διερμηνία. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να μιλάτε υπερβολικά γρήγορα. Επίσης ότι μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μας, στο δίκτυο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και θα υπάρξει μετά και ένα βίντεο για την ακρόαση αυτή. Τώρα, να ζητήσω από την Συπρόεδρο, την κυρία Κάμερβερτ, παρακαλώ, να πει και εκείνη δύο λόγια. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, αγαπητέ ε, κύριε Μπούζεκ, ε, και για τις διευκρινήσεις ε, που δώσατε τόσο σαφώ ω προ το πώ θα τρέξει η σημερινή διαδικασία ακρόαση. Και εγώ, εξ ονόματο τη Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδεία, θα ήθελα να ε, καλωσορίσω θερμά εδώ την οριστήσα Επίτροπο, κυρία Γκαμπριέλ. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή για τον Πολιτισμό και την Παιδεία είναι αρμόδια για το τομέα της πολιτικής οπτικοακουστικών μέσων και ε, τις πολιτισμικές και παιδαγωγικές πτυχές της κοινωνίας της πληροφορίας. Η Επιτροπή είναι ταυτόχρονα ε, γενικά αρμόδια για τα ζητήματα της διατήρησης και της προώθησης πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι βέβαια πάρα πολύ σημαντικά για το συγκεκριμένο ε, χαρτοφυλάκιο και ειδικότερα τα οπτικοακουστικά μέσα και το δημιουργικό τομέα. Η ψηφιακή εποχή μα δίνει πολλέ δυνατότητε, αλλά θέτει και σημαντικέ προσκλήσει. Ω οριστή επίτροπο, αγαπητή κυρία Γκάμπλερ, θα γνωρίζετε βέβαια ότι θα παρακολουθούμε εμεί πάρα πολύ προσεκτικά τι μελλοντικέ εξελίξει, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα βρούμε την κατάλληλη ισορροπία δηλαδή την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στις ε, οικονομικές, τεχνικές και εμπορικές επιταγές αφενός και την ανάγκη να έχουμε να, να διασφαλίσουμε και να προωθήσουμε ε, το πολιτισμικό και ε, δημιουργικό περιεχόμενο αφετέρου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ε, γραπτές απαντήσεις που δώσατε στα ερωτήματα που είχαμε θέσει προκατακτικά ε, και χαίρομαι ε, και με βέβαια ότι θα μας διευκρινίσετε στο πλαίσιο των τριών ουρών που θα ακολουθήσουν τις απόψεις σας για αυτούς το μέσο πολιτικής. Είμαι βέβαια ότι θα απαντηθούν τα κύρια ερωτήματα όλων των επιτροπών στο πλαίσιο αυτής της ακρόασης και αναμένω μεγάλο ενδιαφέρον την πολύ καλή συζήτηση που θα ακολουθήσει και δίνω και πάλι το λόγο στον συμπρόεδρο μου, τον κύριο Μπουζέ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ναι, εγώ θα γυθώ στο πρώτο κομμάτι της συνάντησής μας αυτής, στο 50% των ερωτήσεων λίγο πολύ και η κυρία Κάμερ Βέρτ ως συνπρόεδρος θα αναλάβει όλες τις επόμενες ερωτήσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και εσά που δώσετε τη δυνατότητα στην Επιτροπή Πολιτισμού να συμμετάσχει. Από πλευρά της ε, Ήτρε θεωρούμε και εμείς ότι τα δίκτυα επικοινωνίας, η πληροφορική, η ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων είναι και δικό μας θέμα. Λοιπόν, ας περάσουμε στη συζήτηση. Στην αρχή, όπως είπαμε, θα δώσω το λόγο στην σε επίτροπο για μια παρουσίαση 15 λεπτών. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε Μπούζεκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρία Κάμερβερτ. Πρόεδρε των Επιτροπών ε, Προστασίας του Καταναλωτή, κυρία Σβόμποντα, Πρόεδρε νομικής, ε, Νομικών Υποθέσεων, κύριε Μαρές, και Πρόεδρε της Επιτροπής ε, Δικαιοσύνης Ελευθερίας των Πολιτών, αξιότιμοι συντονιστές και μέλη των επιτροπών αυτών, Ήτρε, Καλτ, Ίμκο, Τζούρι και Λίμπε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα που μπορώ να σα μιλήσω εγώ ως οριστής επίτροπος για το θέμα τη ψηφιακή οικονομία και τη κοινωνία. Ελπίζω ότι σήμερα θα έχουμε μια επικοδομητική συζήτηση για το πώ μπορούμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ψηφιακή ενιαία αγορά μαζί. Υπέρ τη ανταγωνιστικότητα, υπέρ μια Ευρώπη. Ε, με συμμετοχή όλων στην ανάπτυξή της. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε πολλές και πλούσιες ιδέες και θα μπορέσουμε όλοι μαζί να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει η Επιτροπή Γιούγκερ προκειμένου να ελευθερώσουμε όλο το δυναμικό που υπάρχει από την ψηφιακή τεχνολογία. Επιτρέψτε μου όμως πρώτα απ' όλα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. Θέλω να ευχαριστήσω τη βουλγαρική κυβέρνηση που με εμπιστεύτηκε. Αλλιώς δεν θα βρισκόμουν εδώ σήμερα ενώπιό σας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω εσάς, ευρωβουλευτές, για την στήριξη που με έχετε προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν εδώ. Χάρη σε εσά επίσης βρίσκομαι εδώ σήμερα. Βρίσκομαι εδώ λοιπόν ενώπιόν σας για να ζητήσω την εμπιστοσύνη σας για άλλη μια φορά ζητώ να αναλάβω νέες αρμοδιότητες. Και θέλω να ευχαριστήσω και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που και αυτοί με βοήθησαν να ανταποκριθώ στις προκλήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τις χώρες μέλη και το Συμβούλιο επίσης, στο οποίο βρέθηκα συχνά για να διαπραγματευτώ στα πλαίσια των τριμερών διαλόγων. Οι τριμερείς διάλογοι αποτελούν μια ευκαιρία για μας να συμβρεθούμε για να πετύχουμε τους κοινού μας στόχους. Θέλω να ευχαριστήσω και τους Ευρωπαίους πολίτες για την εμπιστοσύνη τους, για τη στήριξή τους σε όλες τις μάχες που έχω δώσει μέχρι σήμερα. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, δεν ήθιστε να κάθετε κανείς εδώ που κάθομαι εγώ αυτή τη στιγμή και να απευθύνεται σε εσά ως οριστής επίτροπος. Αποτελεί προνόμιο όμως, αλλά αποτελεί και πρόκληση και ευκαιρία συνάμα. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν για μένα να συνεχίσω το έργο μου υπέρ των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των Ευρωπαίων πολιτών και να ενισχύσω την παρετέρω ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο στο εσωτερικό όσο και απέναντι στον κόσμο όλο. Είμαι έτοιμη να απαντήσω στις ερωτήσεις σας και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μεταξύ μας υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών. Ποιο, ποια είναι η κύρια πρόκληση που έχουμε σήμερα μπροστά μας και που ενδιαφέρει τους πολίτες είναι η ψηφιακή ενιαία αγορά. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα βασιστώ στην εμπειρία μου για να μπορέσω να βοηθήσω και θα είμαι αποφασιστική για να πετύχω τον στόχο αυτόν. Πρώτα λοιπόν, ε, εμπειρία είχα ως ερευνήτρια στα πλαίσια δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Έτσι λοιπόν θα αντλήσω πόρους για να χρησιμοποιήσω μια καινοτόμο μέθοδο εργασίας στην, ε, για την εξέβρεση λύσεων. Η εμπειρία που είχα μέχρι τώρα με βοήθησε να καταλάβω πόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και οικονομικά την έρευνα προκειμένου να έχουμε στη διάθεσή μας δεδομένα και τα δεδομένα αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλους και να μπορούν όλοι οι Ευρωπαίοι να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Μόνο έτσι θα μπορούμε να βρισκόμαστε στην αιχμή των τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων και έτσι να κατοχυρώσουμε την ευρωπαϊκή αριστεία. Ω πολιτικό λοιπόν που θα παίρνει αποφάσεις πιστεύω ότι πρέπει να δράσουμε και εγώ δεσμεύομαι εδώ να χρησιμοποιήσω ό,τι μέσα μπορώ για να πετύχω ακριβώς αυτό το στόχο. Επιτρέψτε μου επίσης να σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα γιατί έχω και εκεί εμπειρία και από εκεί θα μπορέσω να αντλήσω πόρους. Στη διαδρομή μου λοιπόν είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ με μια πολιτική που στην αρχή δεν ήταν τόσο ελκυστική. Αλλά μετά από τον διάλογο που φρόντισα να υπάρχει, από την ενημέρωση και με πολύ συγκεκριμένα ε, παραδείγματα υπέρ των πολιτών, κατάφερα να πείσω τον κόσμο και να πετύχω πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Πρόκειται για την κοινή γεωργική πολιτική στη Βουλγαρία το 2011. Είχα εκλεγεί τότε μόλις το 2011 και ξεκίνησα μια εκστρατεία πληροφόρησης απέναντι στους αγρότες, οι οποίοι ήταν πολύ σκεπτικιστοί και δεν θέλαν ή δεν είχαν τη δυνατότητα μέχρι τότε να συμμετέχουν σε συζητήσεις για αυτή την πολιτική. Είχα λοιπόν μαζί τους τακτικές ανταλλαγές απόψεων και κατάφερα να τους μεταφέρω επιχειρήματα τα οποία δείχνουν ότι οι πολίτες μπορούν να υποφεληθούν περισσότερο από την πολιτική αυτή για την περίοδο 2014-2020. Θα βασιστώ λοιπόν στην εμπειρία μου αυτή για να χρησιμοποιήσω την ίδια μέθοδο εργασίας. Μια μέθοδο εργασίας που βασίζεται στο διάλογο, στο άνοιγμα και στη συνεργασία. Από εκεί και πέρα, ποια είναι η αποστολή μου. Στην επιστολή που μου απίφθινε ο πρόεδρος Γιούνκερ για την αποστολή μου, αυτή αναφέρεται ρητά. Είναι η διευκόλυνση της ε, έγκρισης και η εκτέλεση των ευρωπαϊκών ε, πολιτικών αποτελεσματικών για να ολοκληρωθεί και να πετύχει η ψηφιακή ενιαία αγορά. Βασίζομαι λοιπόν σε συλλογικό έργο, σε συλλογική δουλειά. Με τον ε, Αντιπρόεδρο Αντσίπ, για παράδειγμα, που είναι υπεύθυνο για την ψηφιακή ενιαία αγορά, και με όλη την ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και τους Ευρωβουλευτές και το Συμβούλιο. Είναι δικιά μας ευθύνη σήμερα να συνεισφέρουμε για να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον τέτοιο που θα επιτρέψει σε όλους τους Ευρωπαίους να υποφεληθούν πλήρως από τις δυνατότητες που δίνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες σήμερα. Τεχνολογίες οι οποίες δεν γνωρίζουν σύνορα. Οπότε τι διαπιστώνουμε σήμερα, δύο χρόνια μετά από την έκκληση που έγινε υπέρ της στρατηγικής για την ψηφιακή ενία αγορά, πρώτα απ' όλα πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι έγινε μια ένα το έργο από τον προκάτοχό μου, τον Επίτροπο Έτιγκερ, σε συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο Αντσίπ. Και τι μου μας δείχνει λοιπόν η στρατηγική αυτή, η οποία αξιολογήθηκε τον Μάιο που μας πέρασε, δείχνει, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ναι, μας μένουν ακόμα πράγματα όπως είναι η ασφάλεια στον κυβερνοχρόνο, η ανάπτυξη, η απασχόληση, ο πολιτισμός, η νεολαία, ε, τα ψηφιακά, οι πολιτικές μας για την ε, εξωτερική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στην Αφρική, η ψηφιοποίηση της βιομηχανίες μας, η ε, συνδεσιμότητα, όλα αυτά τα θέματα παραμένουν πάρα πολύ σημαντικά για όλους μας. Γιατί ναι, το ψηφιακό έχει μια διάσταση που μόνο στον πληθυντικό μπορούμε να την ορίσουμε. Κανένας τομέας δεν μπορεί να εμποδίσει ε, την ψηφιακή εξέλιξη, η οποία επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής μας και κανείς δεν πρέπει να αποκλείεται από αυτήν. Συνεπώς, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι η δικιά μας προστιθέμενη αξία, η ποικιλομορφία και ο συμβιβασμό. Να, τι είναι αυτό που έχουμε να προσφέρουμε. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το καλύτερο παράδειγμα για να δείξουμε τι σημαίνει ένα πραγματικό εργαστήριο ιδεών και τι σημαίνει ποικιλομορφία και συμβασμός. Σήμερα στην Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές συμφερόντων που υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παρά μόνο μέσα από συμβασμούς. Και ακριβώς αυτή τη μέθοδο ανοίγματο και διαλόγου είναι που προτείνω και εγώ για την θητεία μου ως Επίτροπος. Έφτασε η ώρα. Η απάντηση είναι ναι, με ένα μεγάλο ναι. Δύο χρόνια βέβαια θητείας δεν είναι αρκετά. Το αντιλαμβάνομαι. Συνεπώς, τι πρέπει να κάνουμε, ποια είναι η λέξη κλειδί, προτεραιότητες. Η προτεραιότητά μου θα είναι λοιπόν να διασφαλίσω την πλήρη εκτέλεση των πρωτοβουλειών που έχουν ήδη εγκριθεί μέχρι τώρα. Σκοπεύω όμως επίσης να προτείνω και νέες ιδέες. Θα συνεργαστώ με όλους τους επιτρόπους, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το Συμβούλιο και όλους τους ενδιαφερόμενους με έναν ανοιχτό τρόπο, με διαφάνεια, προκειμένου να διασφαλίσω την συνένεση με την συμμετοχή όλων. Ποια είναι η εμβέλεια της ε, ψηφιακής αλλαγής τεράστια. Αποτελεί πηγή τεράστιων ευκαιριών για τον κόσμο. Βοηθάει όμως επίσης να αντιμετωπιστούν και οι μεγάλες σημερινές προκλήσεις. Η ασφάλεια, η υγεία, η φτώχεια, οι ανισότητες, κλιματική αλλαγή. Αυτά είναι όλα. Η ταχύτητα και το βάθος τώρα της αλλαγής οδηγεί σε άλλες μεγάλες προκλήσεις. Έχουμε μια επανάσταση μπροστά μας και πρέπει να φροντίσουμε για αυτήν. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της απώλειας ε, θέσεων απασχόλησης ή των αλλαγών στα μοντέλα δουλειάς μας, πώς θα προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις στις αλλαγές που αφορούν το δικό τους επιχειρηματικό μοντέλο, υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για άντρες και γυναίκες ε, στην ψηφιακή κατάρτιση και στους μισθούς πώς θα διασφαλίσουμε αποτελεσματική ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών στην υγεία, στην διακυβέρνηση, στις μεταφορές και πώς θα φροντίσουμε να υπάρχουν κέρδη και ευκαιρίες για τους πολίτες. Ποιο είναι ο δικός μου χάρτης πορείας θα έχει το στίγμα της απόλυτης αναγκαιότητας για επιτυχή λειτουργία των μέσων που έχουν εγκριθεί από το 2015 και μετά και που εντοπίστηκαν και στην αξιολόγηση στα μέσα του δρόμου. Δηλαδή, κατάργηση του, των τελών roaming ή δυνατότητα μεταφοράς περιεχομένου, η πρωτοβουλία Wi-Fi 14 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δικαιώματα των ε, δημιουργών, η επαναδιάθεση του φάσματος, η υψηλή ταχύτητα σε ευρωζενική συνδεσιμότητα και η εφαρμογή τη συμφωνία του Μαρακέ. Θέλω να υπάρχει επίση καλύτερη συνοχή ανάμεσα στι εσωτερικέ και εξωτερικέ μα πολιτικέ και θα λάβω υπόψη μου και όλε τι κοινωνικέ πτυχέ. Θα προσπαθήσω να πετύχω πολιτικέ συμφωνίε επίση όσον αφορά τον κώδικα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα δικαιώματα των δημιουργών, τη μεταρρύθμιση για το οπτικοακουστικά και το γεωγραφικό αποκλεισμό, κάτι το οποίο δεν δικαιολογείται πια. Θα προτείνω επίση στοχευμένε πρωτοβουλίε στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ξεκινώντας από την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής και θα φροντίσω για επιπλέον μέτρα όσον αφορά τα πρότυπα της ασφάλειας στο κυβερνοχώρο, όπως για παράδειγμα πιστοποίηση και σήμανση. Θα διασφαλίσω επίσης την ασφάλεια όσον αφορά τα δεδομένα ιδιωτικού βίου και ασφάλεια των δεδομένων και συγχρόνως θα διασφαλίσω και ότι τα δικαιώματα τα οποία είναι της Ευρωπαϊκή Ένωση, θα κυκλοφορούν ελεύθερα. Θα δουλέψω λοιπόν πάνω σε όλες αυτές τις πλατφόρμες για δικαιοσύνη, για προσβασιμότητα και για την διάθεση των δεδομένων που έχουν πληρωθεί με δημόσιο χρήμα. Θα δώσω επίσης εξίσου πολύ σημασία στην πρόκληση της ψηφιακής μετατροπής στην ευρωπαϊκή κοινωνία και το κοινωνικό μας μοντέλο. Θα εργαστώ για την ανταγωνιστικότητα, την ηγετική θέση στην τεχνολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα μεγάλα, μεγάλου όγκου δεδομένα, στα σούπερ κομπιούτερ, στην τεχνητή νοημοσύνη και συγχρόνω στα αγωνιστών, για να υπάρξει μια καλή ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα των πολιτών, των επιχειρήσεων και όλων των διαφορομένων, προκειμένου όλοι να μπορέσουν να υποφεληθούν από την ψηφιακή καινοτομία. Ναι, λοιπόν, πράγματι, η τεχνολογία αλλάζει τη ζωή μας. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε, τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε, τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Όμως, ένα είναι ο δρόμος μπροστά μας. Είναι αυτός που δεν μπορεί να παρακάμψει την ενοποίηση. Πρέπει να παραμείνουμε μαζί ενωμένοι και να εργαστούμε για ένα κοινό σκοπό, για το μέλλον της Ευρώπης μας, για το μέλλον των αξιών μας. Ήμουνα μία από εσά όταν είχαμε τις ακροάσεις για τους επιτρόπους ε, της Επιτροπής γιούνκερ. Οπότε θέλω να σας ευχαριστήσω, ε, συνάδελφοι, για τις προσπάθειες που κάνατε μέχρι σήμερα να συντάξετε τις ερωτήσεις. Αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες σας και τις προσδοκίες σας. Επαναλαμβάνω λοιπόν τη δέσμευσή μου όλα αυτά να τα λάβω υπόψη μου σε όλους τους τομείς που έχουν να κάνουν με το τόσο σημαντικό χαρτοφυλάκιό μου. Το μέλλον είναι το πιο σημαντικό από όλα. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν τη στιγμή αυτή για να σας πω ότι θα φροντίσω για την ολοκλήρωση της ψηφιακής αγοράς. Αυτό μπορώ να το πετύχω μόνο με τη δικιά σας ε, τη στήριξη, με τη στήριξη βέβαια και των εμπειρογνωμόνων στις διάφορες γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα βρίσκονται υπό την δική μου ηγεσία οι προσπάθειες πρέπει να είναι κοινέ, γιατί έχουμε και κοινού στόχους, που είναι η προστασία των συμφερόντων των πολιτών μας. Ευχαριστώ. Uh, let us move to the list of... Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Ας περάσουμε τώρα στο κατάλογο των ομιλητών. Θα ήθελα να σας επενθυμίσω ότι έχουμε ένα συν δύο λεπτά και από εκεί και μετά μπορείτε να κάνετε μια επακόλουθη ερώτηση ε, για ένα λεπτό, η οποία πρέπει να απαντηθεί μέσα σε ένα λεπτό. Ξεκινάμε λοιπόν, η κυρία Πέλα Δεκαστήλο. Ε, ε, dear Commissioner Designated. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και αξιότιμη ορθήσα επίτροπε. Καταρχήν να σας πω ότι είναι μεγάλη μας τιμή το γεγονός ότι ήσασταν ένα εξαιρετικό μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τα τελευταία 8 χρόνια. Όπω γνωρίζετε, στην Επιτροπή ΕΙΤΡΕ λαμβανόμαστε τόσο τη βιομηχανία όσο και των ε, τηλεπικοινωνιών και ε, τη ενέργεια αλλά και τη έρευνα και τη καινοτομία. Οπότε, σε ό,τι αφορά σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία τάση για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Πώ μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι όλε οι επιχειρήσει συμπεριλαμβανομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν πρόσβαση σε αυτέ τι τεχνολογίε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Επίτροπο. δύο λεπτά για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Καστελιό, για αυτή την ερώτηση που με οδηγεί ακριβώς στο πυρήνα των προβληματικών που μας ενδιαφέρουν ω Ευρωπαίοι. Πραγματικά τον Απρίλιο του 2016 ευθετήσαμε αυτή την στρατηγική ανακοίνωση που αφορά την βιομηχανία των ψηφιακών επικοινωνιών μέσα σε εξήγηση χόφερ. Σήμερα το διακύβευμα είναι ξεκάθαρο ότι η Ευρώπη έχει σημειώσει επιτυχίες και έχει δυνάμεις. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε ώστε και πάλι να αποτελέσουμε τους ηγέτες επενδύοντας στις βιομηχανίες για μας σημαίνει ότι προετοιμάζουμε το πεδίο ώστε να έχουμε ένα κατάλληλο περιβάλλον που θα επιτρέψει στους μελλοντικού Ευρωπαίους πρωταθλητές παγκόσμιας εμβέλειας να διατηρήσουν το ρόλο τους. Γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να ξεκινήσω από τη σημασία που έχει αυτό το θέμα, ύψιστη δηλαδή στο πολιτικό θεματολόγιο και στη Ρώμη το Μάρτιο αποφασίσαμε την δημιουργία της πλατφόρμας της ψηφιακής βιομηχανίας στην Ευρώπη και επ' αυτού θα επενδύσουμε πολλά και προσπάθειες και πόρους. Δεύτερον, κάτι που είναι εξίσου σημαντικό. Τώρα έχουμε 500 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπονται για την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων. Αυτό μέσω μιας συγκεκριμένης, συγκεκριμένου εγχειρήματο, τα ψηφιακά hubs, η ψηφιακή κόμβη. Είχαμε 150 νέους κόμβους καινοτομία στην Ευρώπη πρόσφατα. Και αυτό ακριβώς είναι το διακύβευμά μας, να μην παραμένει συγκεντρωμένο μόνο σε λίγα σημεία, να είναι διάσπαρτο στην Ευρώπη και να επιτρέψει σε όλους να διαδραματίσουν το ρόλο τους. Γιατί ακριβώς αυτό το κόμβο δεν έχουμε μόνο μεταφορά τεχνολογίας, αλλά αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε πειραματισμό, να έχουμε περισσότερη γνώση και να προωθήσουμε την μηχανία μας. Ευχαριστώ πολύ. Είναι παρακαλώ ένα λεπτό εσείς. Ε, ναι. Σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση της οικονομίας μας, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η σύνδεση, η διασυνδεσιμότητα. Για παράδειγμα, το Wi-Fi for You του Wi-Fi Action Plan, το σχέδιο δράσης, πώς αυτά λοιπόν μπορούν να ε, συμβάλλουν στην ψηφιοποίηση τη Ευρωπαϊκή οικονομίας. Αυτό είναι το ερώτημα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ευχαριστήσα, Πέτρο Ναι, αυτό για μένα είναι μια πρωτοβουλία συμβολική. Γιατί στην προσπαθία μας ψηφιοποίηση των βιομηχανιών θα αναζητήσουμε τους καταλήτες, τους μοχλούς Δηλαδή, κάθε φορά που θα έχουμε μια υπηρεσία, κάθε φορά που θα κάνουμε σύνδεση σε ένα σημείο, θα έχουμε μια αυτόματη σύνδεση και σε άλλα σημεία, ώστε να έχουμε ταυτόχρονα και άλλες υπηρεσίες και μέσω της διασυνδεσιμότητας ακριβώς να προκαλέσουμε αυτό το άνοιγμα του δικτύου. Νομίζω ότι έχουμε ακριβώς ένα εγχείρημα ΣΔΙΤ, όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τη βοήθεια του δημοσίου μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο. Thank you very much, madam. Mr. Dan Nika, your five slot. Ευχαριστούμε ο κύριος Dan Nika ε, και τα πέντε λεπτά για τον διάλογο σας. Ευχαριστώ. Ως οριστής επίτροπος θα κάνετε προτάσεις σε ό,τι αφορά ε, ε, ε, κλήσει για την υποβολή προσφορών είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είτε σε διεθνέ επίπεδο, όπω έγινε και στην περίπτωση τη περιαγωγή ε, του roaming. Δηλαδή, πώ θα διασφαλίσετε ότι οι μεγάλε επιχειρήσει δεν θα αρχίσουν να ουσιαστικά παίρνουν τι περισσότερε από αυτέ τι ε, προκηρύξει για να αντισταθμίσουν τι απώλειε των κερδών του από την περιαγωγή. Επίση, πώ θα αντιμετωπίσετε του αυξημένου κινδύνου τη κυβερνοασφάλεια ως ε, αρμόδια επίτροπος για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία πώς ε, θα προωθήσετε περισσότερο ε, το συντονισμό και την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ, λέω Πρόεδρος. Τρία ερωτήματα θέσατε. Ας ακούσουμε τώρα την απάντηση. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Τάντη για αυτές τις δύο σημαντικές ερωτήσεις. Καταρχάς για τις διεθνείς κλήσεις. Συμφωνούμε για την αρχή ότι η τιμολόγηση δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το κωδικό της χώρας. Αυτό που είναι σημαντικό σήμερα είναι να δούμε ξεκάθαρα ότι υποχωρούν οι, ξα... οι κλήσεις, αντίθετα αυξάνονται οι κλήσεις μέσω εναλλακτικών παρόχων. Η Κομισιόν λοιπόν έχει προτείνει ένα στοιχείο το οποίο κατά την άποψή μου είναι αυτό που βρίσκεται στον πυρήνα αυτού του ζητήματος, δηλαδή ο καθολικός χαρακτήρας παροχής αυτών των υπηρεσιών που θα πρέπει να διασφαλίζουν ακριβώς τη διαθυσμότητα σε όλους τους πολίτες ώστε αυτοί να έχουν δυνατότητα επιλογής. Ελπίζουμε βέβαια και αυτή η τάση για τις αναλλακτικές υπηρεσίες over the top να συνεχιστεί, να περιλάβει τις διεθνείς κλήσεις και να μας επιτρέψει βεβαίως να ασκήσουμε πίεση στις παραδοσιακές υπηρεσίες κλήσεων. Ξέρω ότι υπήρξαν τροπολογίες του Κοινοβουλίου που κατατέθηκαν από αυτού, αυτό είναι τμήμα τη συζήτηση για το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά είναι ξεκάθαρη η Κομισιόν σε σχέση με την προσέγγιση που υιοθέτησε. Εμεί θεωρούμε ότι αυτό διέρχεται από την υπηρεσία καθολικού χαρακτήρα, ώστε να διασφαλίσουμε και να πετύχουμε τιμέ, τιμολόγηση των κλήσεων προσβάσιμε για όλου του πολίτε. και για τι επιθέσει στον κυβερνοχώρο σήμερα είναι ξεκάθαρα ότι ένα από τα διακυβευόμενα που αντιμετωπίζουμε όχι μόνο η βιομηχανία αλλά ολόκληρη η κοινωνία μα, οι δημοκρατικοί μα θεσμοί είναι ακριβώ αυτέ οι απειλέ στον κυβερνοχώρο και πρόσφατα είχαμε εμπειρίε αντίστοιχε. Αυτό τι μα κατέδειξε ότι οι κρίσιμε υποδομέ τη βιομηχανία και η υγεία αυτών των υποδομών στι ε, μεταφορέ πρέπει να προστατεύονται. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σε θέση να έχουμε συγκεκριμένα εργαλεία μέσω σήμανση των προϊόντων, μέσω αδειοδότησης, μέσω καλύτερης επιχειρησιακής δυνατότητας των χωρών μελών να χρησιμοποιούν τους πόρους τους. Εδώ θα σταματήσω. Ευχαριστώ. Κύριε Σαντάνε, το λόγο σε ό,τι αφορά ε, το αγώμα της ε, ε, του e-privacy θεωρείτε πως θα υπάρξει ο κατάλληλος χρόνος προκειμένου να ανταπτυχθεί το κατάλληλο λογισμικό έτσι, και να εφαρμοστεί με το κατάλληλο τρόπο προκειμένου να ανταποκρίνεται στα όσα προβλέπει η σχετική οδηγία για το e-privacy. Ή μήπως θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια παράταση εδώ. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η απάντηση τώρα. Ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση που είναι πολύ σημαντική. Να επενθυμίσω την αρχή που ε, μας επέτρεψε να έχουμε μπροστά μας την πρόταση για την ηλεκτρονική ιδιωτική ζωή. Αν δεν έχουμε το GDPR, το οποίο μας επιτρέπει ακριβώς την προστασία των προσωπικών δεδομένων βάσει του άρθρου 8 της χάρτας, θα έχουμε τον χάρτη της ηλεκτρονικής ιδιωτικής ζωής σε σχέση με τις επικοινωνίες. Γνωρίζω ότι υπάρχουν θέματα για τα οποία θα πρέπει ακόμα βεβαίως να συζητήσουμε. Εξαλλού, η Κομισιόν προτίθεται να το πράξει. Εγώ όμως θα ήθελα να μην ξεχνάμε ποιο είναι ο στόχος που έχουμε θέσει. Σήμερα οι Ευρωπαίοι πολίτες εξέφρασαν ανησυχίες για ασφάλεια για τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι τις συσκευές τους, για να, να προστατεύονται τα δεδομένα τους. Πέρασα το χρόνο μου, σταματάω, η επιδρόμος. Σας ευχαριστούμε. Σαν Εύζεν, του έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα καταρχήν να σας ε, συγχαρώ για το διορισμό σας και αναμένω μια καλή συνεργασία μαζί σας με βάση και την κοινή εμπειρία που είχαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, με βέβαιο ότι θα είστε ένα αντάξιο, ε, μια αντάξη διάδοχο του κυρίου Ότιγκερ. Τώρα, ε, θα ήθελα να σα ρωτήσω κάτι σχετικά την ενίσχυση του Μπέρεκ, του Ευρωπαϊκών Θρηστικών Αρχών για τις ηλεκτρονικές ε, επικοινωνίες. Θα ήσασταν διατεθειμένοι να ε, τροποποιήσετε ε, την πρόταση της Επιτροπής σε σχέση με το ΜΠΕΡΕΚ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστής Επιτροπός. ευχαριστώ πολύ το, Βουλός και αυτή την ερώτηση. Σέβομαι πολύ του δουλειά ως εισηγητή και γνωρίζω την ανάγκη περισσότερη συζήτηση επειδή σήμερα υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τις θέσεις των θεσμικών οργάνων. Για μένα είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ποιος είναι ο στόχος μας. Το ΜΠΕΡΕΚ έχει ένα σημαντικό ρόλο ακριβώς για να επιφέρουμε κάποια σαφήνεια, κάποια συνάφεια, για να έχουμε ένα ευρωπαϊκό όραμα. Πώς αυτό το στον τομέα μπορούμε να πετύχουμε κοινού στόχου με όσο πιο δομημένο τρόπο γίνεται. Είναι ξεκάθαρο ότι το ΜΠΕΡΕΚ έχει διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο πρόσφατα στην περιεγωγή και στην ουδετερότητα στο διαδίκτυο. Αν δούμε το γραφείο του ΜΠΕΡΕΚ, είναι η πιο μικρή υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 28 υπαλλήλους. Ταυτόχρονα όμως ξέρουμε το πώς μια υπηρεσία δουλεύει, με ποιο φόρτο δουλεύει εργασίες και πώς συνεργάζεται αυτή η υπηρεσία με τους εθνικούς ρυθμιστές. Από για μένα σήμερα, το ζήτημα που τίθεται είναι κατά πόσο θα πρέπει να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα αυτή η δομή. Γι' αυτό ακριβώς θα συνεχίσω σε βάθος τις συζητήσεις με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ώστε να εντοπίσω ένα κοινό παρανομαστή που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε. Γιατί αυτό θέλουμε. Θα προχωρήσουμε όσο μπορούμε. Αλλά ξέρουμε ότι στο ψηφιακό κόσμο δεν έχουμε πολύ χρόνο. Οπότε όλοι θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες και από αυτού θα δεσμευτώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να θέσετε επακόλουθο ερώτημα. Ναι, πολύ σύντομα. Πρώτα καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά ε, την κυρία Γκάβριελ για αυτήν την καλά θεμελιωμένη απάντηση. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω και το εξή. Ο Μπέρεκ ε, βασίζεται στο κώδικα. Οπότε, ε, ποιο θεωρείτε πως είναι το πρόβλημα εδώ σε σχέση με το φάσμα. Γιατί Είπατε σωστά ότι χρειάζεται να διασφαλίσουμε τον ε, κατάλληλο συντονισμό αλλά και την εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από την άλλη όμως ε, πλευρά θα πρέπει ε, να επιτρέπουμε στα κράτη-μέρη να αναλαμβάνουν τα καθήκοντα που τους αναλογούν. Δηλαδή εδώ βέβαια έχουμε να κάνουμε και πάρα πολύ με ζητήματα ανταγωνισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Κύριε Έχω ένα λεπτό στα θέση μου, έτσι, για το φάσμα. Αυτό σχετίζεται άμεσα με την πέμπτη γενιά και τη συνδεσιμότητα. Η πέμπτη γενιά θα μας επιτρέψει να αποτελέσουμε εμείς την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη όλων. Ξέρω ότι όταν μιλάμε για κατανομή φάσματος, αμέσως ανακέπτουν διαφορές όσον αφορά τη θέση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Κομισιόν. Εγώ προσωπικά πιστεύω θα πρέπει να πάρουμε θέση και θα πρέπει να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό. Αυτός είναι ο στόχος μας σήμερα. Αν αυτό βέβαια διέρχεται από περισσότερες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε ας μην ξεχνάμε ότι για μας σήμερα αυτό αποτελεί μια ευκαιρία. Και ευχαρίστως να ακούσω την θέση των χωρομελών και του Συμβουλίου όμως για την κατανομή του φάσματος πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα όταν μιλάμε για ευρωπαϊκή προσέγγιση να συνοδεύονται τα λόγια από πράξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τα επόμενα πέντε λεπτά ε, στο συνάδελφο Κάλια Κάλλας. Στη συνάδελφο Κάλλας. Ναι, βρίσκομαι εδώ. Ε, νομίζω πως ε, το κλειδί για να επιτύχουμε στην ε, ψηφιακή οικονομία και στην ψηφιακή κοινωνία είναι εμπιστοσύνη. Δηλαδή αν απολεστεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον τότε είναι πολύ δύσκολο να την ανακτήσουμε. Ωστόσο βλέπουμε όλο ένα και περισσότερες εθνικές κυβερνήσεις να μιλούν για την πάυση της κρυπτογράφησης των επικοινωνιών γιατί θεωρούν πως θα παίξει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Οπότε το ερώτημά μου προς εσά είναι το εξής. Θεωρείτε πως είναι αναγκαίο να διατηρηθεί, να διασφαλιστεί τη κρυπτογράφηση έτσι ώστε να παραμείνει η εμπιστοσύνη από την πλευρά των καταναλωτών ότι οι επικοινωνίες τους είναι προστατευμένες. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και η Οστήσια Επίτροπος τώρα μπορεί να απαντήσει. Να απαντήσω όσο πιο απλά γίνεται. Σήμερα είναι σημαντικό να έχουμε την κρυπτογράφηση ως εγγύηση για την ασφάλεια χωρίς να υπάρχουν πιθανότητες παράκαμψης backdoor. Υπήρξαν ήδη πρωτοβουλίε των χωρών που χρησιμοποίησαν την αποκωδικοποίηση της κρυπτογράφησης και είδαμε ποια αποτελέσματα είχαμε. Είναι λοιπόν ώρα να προχωρήσουμε γιατί η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη των πολιτών θα ανακύψει από μια σειρά μέτρων. Αλλά αυτή, αυτό ακριβώς είναι η αρχή για την οποία προτείνω ακριβώς να πάμε προς την ίδια κατεύθυνση. Okay, thank you very much, madam. Madam Kai. Ευχαριστούμε. Τι έκαλες, είστε πάλι. Ναι, έχω ερώτημα και γίνεται λόγος ε, για την νομική, αν θέλετε, πρόσβαση σε κρυπτογραφημένες ε, πληροφορίες, ε, κάτι που ενδεχομένως από τεχνικής άποψης να μην είναι καν δυνατό, αλλά άρα μας λέτε ότι δεν θα προβλεφθεί μια τέτοια νομικά προβλεπόμενη πρόσβαση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Γκάμπλερ, να απαντήσει. Ναι, η νομική πρόσβαση μπορεί να γίνει μόνο υπό πολύ αυστηρές συνθήκες, όπως και για άλλα νομικά ζητήματα όταν μόνο έχουμε να κάνουμε θέματα εθνικής ασφάλειας Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να προσέχουμε ώστε να έχουμε συνάφεια με άλλες νομοθετικές διατάξεις που διαθέτουμε αλλά και ταυτόχρονα να επιβεβαιώνουμε κάποιες αρχές γενικές ξεκάθαρα. Πρέπει να δίνουμε και τη δυνατότητα στα όργανά μας, στους θεσμούς μας να προχωρήσουν Πρέπει όμως να προσέχουμε ώστε αυτά τα εργαλεία να μην χρησιμοποιούνται από άλλους για στόχους που δεν είναι οι ίδιοι θετικοί στόχοι που έχουμε εμείς κατά νου. Thank you very much. Next time slot for... Σας ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο πεντάλεπτο για την κυρία Μαρίζα Ματίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ στα αριστερά σας είμαι. Αγαπητοί σα Επίτροπε, καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι πραγματικά ήταν πολύ ευχάριστη εμπειρία ε, της συνεργασίας μου μαζί σας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και ε, σε ό,τι αφορά τώρα τα γραπτά ερωτήματα που σας, θέσατε, σας θέσαμε, τις απαντήσεις σας αναφερθήκατε στην ε, δυνατότητα υποβολής νέων νομοθετικών προτάσεων σε διάφορους τομείς σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τις επιγραμμικές πλατφόρμες, τις online πλατφόρμες και τις σχετικές επιχειρήσεις. Εδώ πρόκειται για ένα πολύ ε, σημαντικό ζήτημα, ενώ ελέφαντα, αν θέλετε, μέσα στο δωμάτιο μα απασχολούν πάρα πολύ αυτά τα ζητήματα και είναι αμφιλεγόμενα. Αν θέλετε, δηλαδή το, ε, το Airbnb, η Uber ή άλλου είδου τέτοιε πλατφόρμε, πάρα πολύ γνωστέ. Οπότε θα ήθελα να σα ρωτήσω ε, τι προτίθεστε να κάνετε σε, αυτόν, ε, σε αυτούς τους τομείς σε σχέση με αυτές τις πλατφόρμες, ε, στο κανονιστικό επίπεδο και τι είδους κανονιστική πρόταση ενδεχομένως θα είχατε κατά νου, γιατί μπορεί να είναι πολύ διαφοροποιημένες. Ε, θα θεωρούνται δηλαδή υπηρεσίες παρεχόμενες, πώς θα αντιμετωπίζονται σχετικέ επιχειρήσεις, τι προτίθεστε να κάνετε σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο κύριε Καμπρί Ευχαριστώ κυρία Ματίας. Ανταποδίδω αυτό που είπατε για την συνεργασία. Αυτή την ε, ποικιλία πλατφορμών πρέπει να τη διατηρήσουμε γιατί αποτελούν πηγή καινοτομία. Έχουν διαδραματίσει ένα θετικό ρόλο αυτές οι πλατφόρμες στο τωρινό οικονομικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα όμως, για να δώσουμε ένα παράδειγμα το τι μπορούμε να κάνουμε όταν έχουμε πρόβλημα, γιατί αυτή είναι και η προσέγγιση της Κομισιόν και την αναφέραμε στην ανακοίνωση για τις πλατφόρμες ξεκάθαρα ότι εδώ δεν θέλουμε να υπερνομοθετήσουμε. Όταν όμως έχουμε διαπιστώσει ένα πρόβλημα, τότε κάνουμε προσαρμογές και διορθώσεις. Και επιβεβαιώνω ότι θα υπάρξει μία πρωτοβουλία για τις αθέμητες πρωτοβουλίες μεταξύ πλατφορμών και των επιχειρήσεων που ζημιώνονται από αυτό τον ανταγωνισμό μεταξύ των πλατφορμών. Γιατί είδαμε ότι όντως αυτό υπάρχει χωρίς καμία δικαιολογία οι επιχειρήσεις αποτρέπονται από την πρόσβαση στα δεδομένα των πελατών τους και αυτό ζημιώνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε σήμερα θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι μπορούμε να προτείνουμε για να δώσουμε λύση σε αυτή την κατάσταση. Αλλά βεβαίως προσπαθώντας να διαφυλάξουμε πάντοτε το δικαίωμα του ανταγωνισμού γιατί γνωρίζουμε ότι είμαστε ακριβώς στο όριο. Ξέρουμε ότι αυτές οι αθέμετες πρακτικές δεν γίνεται να τις δεχτούμε. Θέλουμε να στείλουμε λοιπόν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι θέλουμε να υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο θα μας επιτρέπει να έχουμε τις καλύτερες συνθήκες για όλους. Αλλά μέσω ακριβώς και των κανονισμών θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Αυτό βέβαια δεν θα θέτει ένα αμφιβόλο την ελευθερία των πλατφορμών ακριβώς όταν έχουμε κάνουμε με καινοτομία μέσω ακριβώς της οποίας έρχεται το νέο πρότυπο ε, ανταγωνιστικής επιχείρησης. Σας ευχαριστώ πάλι και πάλι σε ό,τι αφορά τις ε, online πλατφόρμες. Αναφερθήκατε σε κάτι σημαντικό, δηλαδή την ελευθερία της έκφρασης, ε, Πράγματι, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια σειρά από διαφορετικούς ε, τομείς, δηλαδή τις πλατφόρμες, τις επιχειρήσεις, ε, ε, ένας όλος τρόπος μέσα τον οποίο μπορούν να εφραστούν οι πολίτες μας. Και ακριβώς εδώ εντάσσονται και online πλατφόρμες. Και εδώ τίθεται και βέβαια και το ερώτημα της online ελευθερίας της έκφρασης και της λογοκρισίας. Δηλαδή, εάν αυτές οι πλατφόρμες περιέχουν βαράνομα περιεχόμενα, ή αθέμητο περιεχόμενο γενικότερα, τίθεται και πάντοτε αυτό το ερώτημα, δηλαδή ανάμεσα στο πώ θα υπάρξει ρύθμιση μεταξύ ελευθερία τη έκφραση και λογοκρισία. Οπότε θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η δική σα ε, άποψη, πώ μπορείτε να αντιμετωπίσετε ε, αυτά τα ζητήματα που είναι ιδιαίτερα αμφιλογόμενα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ευχαριστή Επίτροπο να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ, επιτροπο να απαντησει Ματίας, για τη δεύτερη ερώτηση. Πράγματι, οι πλατφόρμες είναι ένα από, ένα από τα πιο καινοτόμα εργαλεία για την ελευθερία της έκφρασης και της ελευθερίας. Έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν. Και η πλειοψηφία του περιεχομένου που βρίσκεται στις πλατφόρμες αυτές είναι νόμιμο. Και σήμερα ακριβώς επιβεβαιώνουμε την βούλησή μας να συνεργαστούμε με αυτές τις πλατφόρμες ώστε το ταχύτερο δυνατόν να ακυρώσουμε το παράνομο περιεχόμενο. Βλέπουμε σήμερα και άλλα φαινόμενα στην κοινωνία μας, η άνοδος της τρομοκρατίας. Οπότε θεωρώ ότι ήδη διαθέτουμε ένα οικονομικό, ένα νομικό συγγνώμη εργαλείο, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντικό να εργαστούμε πάνω σε θελοντικά, σε θελούσια μέτρα, ώστε να έχουμε τα κατάλληλα αποτελέσματα. έχουμε συμφωνία με τέσσερις μεγάλες πλατφόρμες, Twitter, Microsoft, Facebook και Viber, που μας επέτρεψε να προχωρήσουμε γιατί, γιατί αφαιρέθηκε μεγάλο ποσοστό παράνομο περιεχομένου. Οπότε πρέπει να συνεχίσουμε το διάλογο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις σας. Ε, το επόμενο πεντάλεπτο τώρα για την κυρία Χέλγα ναι. Τρούπερ θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα του ονομαζόμενου value gap, δηλαδή τη στρέβωση της αγοράς που προκαλείται από το γεγονός ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες ε, προσφέρουν ε, κάποιες φορές δωρεάν ε, περιεχόμενο. Ειδικότερα περιεχόμενο που είναι προστατευόμενο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οπότε εσείς ως οριστήσα επίτροπος θα θέλετε να δημιουργήσετε μια γενικότερη ευθύνη σε ό,τι αφορά ακριβώς την online διαβίβαση αυτών των έργων και θεωρείτε πως θα πρέπει να γίνεται εκ των προτέρων έλεγχος σχετικών τεχνολογιών, ε, ε, κοινή χρήση σχετικών δεδομένων. Θεωρείτε δηλαδή ε, πω το σημερινό κανονιστικό πλαίσιο μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την κατάσταση χωρί να χρειαστεί να αναθεωρηθεί η ισχύουσα οδηγία σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, η κυρία Κάμπριλ τώρα να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Τρόπελ για αυτή την τόσο σημαντική ερώτηση. Παρακολουθώ τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο με μεγάλη προσοχή όταν μιλάμε για αυτό το value gap. Σήμερα ο στόχος της Κομισιόν είναι ξεκάθαρος. Να δώσουμε τη δυνατότητα στους δημιουργούς μέσω του περιεχομένου να αποφεληθούν από αυτή την διανομή. Για μένα σημαντικό σήμερα αυτό, γιατί τα πραγματικά δικαιώματα χωρίς ε, σεβασμό, χωρίς τήρησή τους και εφαρμογή τους, δεν ε, βοηθούν τους δημιουργούς. Οπότε θα πρέπει να δούμε ακριβώς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους δημιουργούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό νομίζω. Βλέποντας την πρόταση, θα δούμε ότι αφορά τις πλατφόρμες όταν έχουμε μια κριτική μάζα περιεχομένου στις πλατφόρμες. Για μένα αυτό που είναι σημαντικό είναι να ζητάμε την άδεια του δημιουργού και να έχουμε δυνατότητα να παρανεύουμε. Θεωρώ ότι όλα αυτά εδώ ακριβώς βρίσκονται. Δηλαδή, να θέσουμε πρώτον των ευθυνών τους, τους δημιουργούς που βρίσκονται στο ψηφιακό κόσμο σήμερα, αλλά να τους θέσουμε πρώτο τους επίσης για να συμβάλλουν πλήρως ώστε να υπάρχει ακριβώς πνευματική δημιουργία. Και αυτή η πνευματική δημιουργία ακριβώς διέρχεται από την αμοιβή με το σωστό τρόπο των δημιουργών. Εγώ λοιπόν θα συνεχίσω να παρακολουθώ με προσοχή τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο, το άρθρο 13 αυτού τόσο σημαντικού κειμένου. Για μένα το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Να δώσουμε τα μέσα στους δημιουργού μας, ώστε να δημιουργούν και να θέσουμε τους υπόλοιπους ευλεκόμενους πρώτων ευθυνών τους για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Παρακολουθώ ναι, σε ό,τι αφορά τη συνθήκη του Μαρακέσα, ε, να πούμε ότι υπάρχει μια περιεκτική συμφωνία την οποία λάβαμε το Μάιο. Οπότε θα ήθελα να ακούσω λίγα περισσότερα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία κύρωση από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να προωθήσουμε τι σχετικέ προσπάθειε χωρί να υπάρχουν περαιτέρω καθυστερήσει και προκειμένου να προωθηθεί και περισσότερο η προστασία των σχετικών δικαιωμάτων των ε, βιβλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτή. Οπότε, ε, ε, ε, κύρωση, μπορείτε να μου βεβαιώσετε ότι θα λάβει η χώρα το Σεπτέμβριο επί την Εστονική Προεδρία. Ευχαριστούμε. Ευθύς Επίτροπος. Κύριε Τροπέλ, θα έλεγα ότι ως Ευρωβουλευτής συχνά βρισκόμουν σε αυτές τις καταστάσεις που είχαν να κάνουν με το Συμβούλιο και τη στάση του. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει εμείς να αποδεχθούμε αυτές τις καταστάσεις. Αν λοιπόν εγώ οριστώ στη θέση του Επιτρόπου, αυτό θα είναι από τα θέματα για τα οποία θα δείσω την μεγαλύτερη ευαισθησία ακριβώ για την υλοποίησή του. Γιατί ήδη έχουμε χάσει πολύ χρόνο. Το δικαστήριο είπε ότι το θέμα είναι αρμοδιότητα της Ένωσης, οπότε πολύ ωραία, ώρα να προχωρήσουμε. Thank um, Σας ευχαριστούμε πολύ για την απάντησή σας. Επόμενο πεντάλεπτο, κύριος Μάρκο Ζούλο. Ευχαριστώ την Επιτρόπο. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Γεια σας. Να θέσω κάτι γνωστό, το οποίο όμως δεν έχουμε προσεγγίσει επαρκώς στην Ευρώπη. Η φορολόγηση των κολοσσών από τις ψηφιακές επιχειρήσεις. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η φορολογική αρμοδιότητα είναι εθνική, αλλά στην Ένωση για θέματα ανταγωνισμού θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ίσου ανταγωνισμού, αποτρέποντα ακριβώ τον του ανταγωνισμού, προστατεύοντα του καταναλωτέ. Να ρωτήσω λοιπόν την ε, Επίτροπο, στην πρόταση για τα ψηφιακά που θα βγει φέτο, οι επιχειρήσει οι οποίε ε, προσφέρουν υπηρεσίε συγκρίσιμε με αυτές που προσφέρουν οι επιχειρήσει τη ε, πραγματική οικονομίας θα πρέπει να φορολογούνται στην χώρα μέλο όπου λαμβάνει η χώρα η οικονομική δραστηριότητα και όπου, από την οποία προέρχονται ακριβώς τα κέρδη. Έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο. Κύριε Πίτροπε, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Ζουλό για αυτή τη σημαντική ερώτηση αλλά και πολύ ευρεία γιατί αφορά θέματα των εσωτερικών μας πολιτικών, δηλαδή πολιτικές ανταγωνισμού, αλλά και εξωτερικές πτυχές. Καταρχάς, είναι ξεκάθαρο ότι οι πλατφόρμες δεν είναι υπεράνω του νόμου. Οι κανόνες που υπάρχουν για όλους θα πρέπει να τηρούνται, να είναι σεβαστοί. Εξάλλου, αυτό ήδη συμβαίνει για τις πλατφόρμες που δρούν στην επικράτεια της Ένωσης. Και στη συνέχεια θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές υποθέσεις. Ήδη η Κομισιόν απέδειξε μέσω τη Επιτρόπου Βεστάγκερ και τη γενική Διεύθυνση για τον Ανταγωνισμό ότι όταν έχουμε περιπτώσεις όπως η Apple ή η Starbucks μπορούμε να αντιδράσουμε, δηλαδή να προασπίσουμε τις πραγματικές δραστηριότητες των πλατφορμών όπως έχουν δηλωθεί. Εξάλλου θα πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς και ποια είναι και η δυσκολία με τις πλατφόρμες. Καμιά φορά είναι δύσκολο να αποφασίσουμε να δούμε ποια είναι η σχέση όσον αφορά τη δημιουργία αξίας, γιατί μιλάμε για εμπλεκόμενους, ενδιαφερόμενους που βασίζονται σε μια ποικιλία πηγών. Οπότε εδώ θα πρέπει ακριβώς να δούμε τι θα γίνει με τη συζήτηση που αφορά τη φορολογία αυτών των επιχειρήσεων. Εξάλλου αναφερθήκατε και σε κάτι άλλο σημαντικό, το level Playfield, δηλαδή την ισοτιμία θα πρέπει να έχουμε κανόνες ισότιμους για ισότιμες υπηρεσίες. Η αρχή αυτή υπάρχει σήμερα. Τώρα κατά πόσο αυτό θα περάσει μέσω από νομοθετικά εργαλεία δεν ξέρω. Έχουμε πάντως τα εργαλεία τα απαραίτητα στη διάθεσή μας και μελέτη δικτύπου αλλά και διαβούλευση ώστε να αναζητήσουμε όλα τα απαραίτητα επιχειρήματα που μας ζητούνται. Θα πρέπει όμως να κατανοήσουμε επίσης ότι θα πρέπει να αντιδράσουμε μέσω συνεργασίας, μέσω εθελοντικών μέτρων για να συνεργαστούμε ακριβώς με αυτές τις πλατφόρμες. Για μένα σήμερα είναι ένα θέμα ισορροπίας, δηλαδή οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να παραφέρονται σήμερα. Θα πρέπει εμείς οι ίδιοι ως Ευρωπαίοι να δούμε πώς ακριβώς θα μπορούσαμε να είμαστε πρωτοπόροι σε θέματα νομοθετικού πλαισίου ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Επόμενος ομιλητής. Όχι, ο ίδιος συνάδελφος συνέχεια στην ερώτηση του δευτερολογία. Νομίζω, λέει ο κύριος Τσούλο, ότι η καλύτερη κατανομή των φόρων θα μπορούσε ακριβώς να βοηθήσει πολλές startup επιχειρήσεις στην Ευρώπη, όπως ακριβώς συμβαίνει στην Αμερική θα ήθελα να ρωτήσω στην αεροναυτική τη δεκαετία του 70 δημιουργήθηκε ακριβώς το εγχείρημα της Έρμπας που κατάφερε να ανταγωνιστεί τους Αμερικανούς. Προβλέπεται να υπάρξουν ανάλογα εγχειρήματα στην ψηφιακή οικονομία. Θα μπορούσαν να προβλέψουν επίσης και την ύπαρξη μιας μηχανής αναζήτησης ευρωπαϊκής. Κύριε Επίτροπε, παρακαλώ. Συμφωνώ κύριε Τζούλο με την ανάλυση σας για την αδυναμία αυτή τη στιγμή που παρουσιάζουν οι ευρωπαϊκές ψηφιακές πλατφόρμες. Είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Αυτό όμως θα πρέπει να μας δώσει δύναμη ακριβώς για να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε σήμερα. Και γι' αυτό ακριβώς επανέρχομαι στην αρχική μας αξία, δηλαδή να έχουμε ένα περιβάλλον κανονιστικό το οποίο θα προωθεί την καινοτομία και την έρευνα, συμπεριλαμβανομένων και των startups. Τώρα για την μηχανή αναζήτηση στην Ευρωπαϊκή, μια Ευρωπαϊκή Google, νομίζω ότι είναι σημαντικό για μα να επενδύσουμε σε τομεί κλειδί στον τομέα τη έρευνα, κάτι το οποίο θα μα επιτρέψει να αξιοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά μας πλεονεκτήματα. Ένα παράδειγμα είναι οι μηχανικές πλατφόρμες. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η απαραίτητες επενδύσεις σε υπολογισμούς, υπολογιστικές μηχανές υψηλής αξίας. Θα μπορούσαμε λοιπόν με αυτούς τους τρόπους να δώσουμε στους πολίτες συγκεκριμένες λύσει λύσεις όσον αφορά την πρόληψη των ασθενειών και σε άλλους τομείς. Σήμερα αυτό που θέλουμε είναι πραγματικά η Ευρώπη να παρέχει τη δυνατότητα χρήσης αυτού του ασφαλούς περιβάλλοντος που θα ευνοεί όλες τις start-up τις επιχειρήσεις, ώστε ακριβώς η Ευρώπη να γίνει ένας πρωταγωνιστής όσον αφορά την πρόσπιση του ψηφιακού. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος των ε, ερωταπαντήσεων. Πριν περάσουμε στο δεύτερο τμήμα, θα ήθελα, παρακαλώ, να μεταφέρω την ε, ευθύνη για την Προεδρία πια στην ε, κυρία Πέτρα Κάμεροβερτ. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. Λοιπόν, έχετε και το λόγο και όχι μόνο για να ηγηθείτε. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Μπούζεκ. Ε, και εγώ θα συνεχίσω να είμαι πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά του ε, χρόνου ομιλία και δίνω τώρα το λόγο στην ε, συνάδελφο Σαμπινέα Φεχάιν. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γκάμπριελ. Και η Ευρωπαϊκή και το Κοινοβούλιο θέλουν να προωθήσουν τον πολιτισμό και την ποικιλομορφία. Από ό,τι βλέπω, ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα και των καταναλωτών και των δημιουργών είναι να υπάρχει σταθερότητα στην κατάσταση αυτή, προωθώντας και άλλους πυλώνες ε, της οικονομίας, το διαδίκτυο και τις προϋποθέσεις για την ψηφιακή τεχνολογία. Βέβαια όλο και περισσότερο έργα παράνομα βρίσκονται στο διαδίκτυο χωρίς την άδεια και χωρίς την οικονομική αντιστάθμιση. Εσείς θα υιοθετήσετε επιπλέον μέτρα πέρα από αυτά τα οποία ήδη ισχύουν για να καλυφθεί αυτό το χάσμα και να πάψει πια αυτή η πειρατεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστούμε. Η οριστής επίτροπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Θέλω να το πω ε, ευθύ εξ αρχής, ότι αυτή η πολιτισμική πολυμορφία είναι πραγματικά στην καρδιά μου. Οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες στην Ευρώπη πρέπει να διατηρηθούν. Και είναι πολύ σημαντικό επίσης τα προστατευμένα έργα από τα δικαιώματα του δημιουργού να είναι έργα τα οποία να μπορούν να αποφεληθούν από την ψηφιακή τεχνολογία, συγχρόνως όμως να εφαρμόζουν τις αρχές που θέλουν οι χώρες μέλη, αλλά υπό την ευρωπαϊκή αιγίδα. Σήμερα ξέρω ότι έχουμε ήδη μία πρόταση, αλλά είναι πολύ σημαντικό μαζί με τους δημιουργούς από κοινού να δουλέψουμε για να υποστηρίξουμε τα δικαιώματά τους. Αυτό θα γίνει μέσα από την πρόθεση ευρωπαϊκών έργων. Είναι κεφάλαιο της Ευρώπης αυτό και ξέρουμε ότι συμπεριλαμβάνεται στην τρέχουσα νομοθεσία. Ξέρω ότι εδώ υπάρχουν κάποιες διαφορές ανάμεσα στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των άλλων θεσμικών οργάνων, αλλά για μένα εδώ αυτό που έχει σημασία είναι να υποστηρίξουμε μια αρχή, προκειμένου οι δημιουργοί μας να προβάλλονται και να εποφελούνται επίσης από μια καλύτερη κατανομή. Και αυτό γίνεται και μέσα από τη χρηματοδότηση. Και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που θέλω να φροντίσω ώστε να μπορούν οι δημιουργοί με κάθε ελευθερία να δημιουργούν. Τώρα, για την καταπολέμηση της πειρατείας, την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου και τη δυνατότητα που πρέπει να έχει ο δημιουργός όταν βλέπει ότι χωρίς την αδειά του κυκλοφορεί το έργο του, ναι, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε. Υπάρχει συμπληρωματική ερώτηση. Παρακαλώ. θα ήθελα να θέσω ένα επακόλουθο ερώτημα ως προς το ποιο ρόλο μπορούν να παίξουν εδώ οι online πλατφόρμες. Έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών κανονισμών, χωρίς όμως ε, τελικά κανένας από αυτούς να ταξινομεί ξεκάθαρα τις εν λόγω ε, αυτές ε, πλατφόρμες και να θέτει συγκεκριμένους περιορισμούς. Οπότε το ερώτημά μου είναι, έχετε προβλέψει κάτι συμπληρωματικό δηλαδή έναν τρόπο ρύθμισης αυτών των ε, πλατφορμών έτσι ώστε να αποφύγουμε αυτήν την ε, νομική ασάφεια που ε, ισχύει σήμερα και που τους επιτρέπει ενίοτε να ακριβώς καταστατηγούν τους νόμους. Ίσως δηλαδή θα μπορούσε να υπάρξει ένα συγκεκριμένο ορισμός αυτού του είδους των υπηρεσιών ακριβώς προκειμένου να διασφαλίσουμε εδώ και σαφήνεια. Ευχαριστούμε για να απαντήσει η κυρία Κάμπριελ. Εκτός μικροφώνου. Αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες σας για το ρόλο των πλατφόρμων. Ναι. Σε αυτά τα πλαίσια σήμερα ο ρόλος αυτός πρέπει να καθοριστεί πιο συγκεκριμένα. Αλλά όπως έχω ήδη πει, αυτό δεν θα γίνει με υπερβολική ρύθμιση. Έχουμε την αρχή της περιορισμένης ευθύνης, έτσι όπως καθορίστηκε από την Οδηγία για το Εμπόριο. Ξέρουμε σήμερα ότι είναι πολύ σημαντικό οι πλατφόρμες αυτές να κάνουν την δουλειά που πρέπει να κάνουν όταν ενημερώνονται ότι πρόκειται για παράνομο περιεχόμενο, όταν ενημερωθούν ότι πρόκειται για καταχρήσεις και πρέπει εκείνες να αναλαμβάνουν δράση. Πιστεύω επίσης ότι στα πλαίσια του διαλόγου που έχουμε με τις πλατφόρμες υπάρχει και περιθώριο για θελοντική βάση πρέπει να συνεργαστούν περισσότερο εδώ μαζί τους, ώστε τα μέτρα αυτά που μπορούν να παίρνουν σε θελοντική βάση να προέρχονται από ένα διάλογο που κάνουμε μαζί τους και να επιτρέψουν και καινοτόμα μέσα στη διάθεσή μας. Ευχαριστούμε πολύ. Η Σίλβια Κώστα έχει το λόγο. Θα μιλήσω τελικά, οπότε βάλτε τα ακουστικά σα παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε τις ευχές μου στην Επίτροπο. Ακούσαμε ότι τις αμμοδιότητες είναι η οικονομία και η κοινωνία, οι ψηφιακές. Αλλά νομίζω ότι ελάχιστα έχει αναπτυχθεί η εκπαιδευτική διάσταση. Γίνεται ακόμα συζήτηση για το χάσμα και για τη δυνατότητα δημιουργίας πλατφορμών για σχολεία και πανεπιστήμια, αλλά επίσης μιλάμε και για τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, ιδιαίτερα για τους ανηλίκους. Πώς ε, προτίθεστε να δράσετε σε αυτόν τον τόσο σημαντικό πυλώνα για μας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κώστα, κύριε Γκάμπριλ. Ευχαριστώ κύριε Κώστα, γιατί μου επιτρέπει αυτό να έρθω σε ένα από τα θέματα που θεωρώ πιο σημαντικά. Όπως είπα, η ψηφιακή μετατροπή ε, πρέπει να έχει σαν κέντρο το πολίτη, να υποφεληθεί από αυτήν ο πολίτης δηλαδή. Ακούμε ότι κάποιες θέσεις απασχόλησης θα εξαφανιστούν, κάποιες άλλες θα εμφανιστούν. Το βέβαιο είναι ότι οι περισσότερες θέσεις απασχόλησης θα αλλάξουν, θα τροποποιηθούν. Οπότε το θέμα δεν είναι πού θα χαθούν και πού θα επανεμφανιστούν θέσεις απασχόλησης. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνοδεύσουμε τους πολίτες σε αυτήν την ψηφιακή αλλαγή να δούμε ποιες είναι οι ψηφιακές ικανότητες. Και εδώ δεν μιλάμε μόνο για τους νέους, μιλάμε και για τους ενήλικες, μιλάμε για τους ευάλωτους, υπάρχουν οι, τα άτομα με αναπηρίες. Γι' αυτό η πρωτοβουλία που θα υποστηρίξω είναι αυτή ώστε οι νέοι στην Ευρώπη να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τετράμινες, πεντάμινες εκπαιδεύσεις στα ψηφιακά. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα. Εσείς είσαστε από την Ιταλία και έχετε πάρα πολλά παραδείγματα. Γιατί να μην κάνουμε όπως έχει κάνει και η Ιταλία ε, για την εγγύηση για τους νέους. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους νέους, ώστε με ευρωπαϊκά χρήματα να φανεί η ευρωπαϊκή αξία μιας εμπειρίας από την οποία όλοι έχουν επωφεληθούν. Και θα επικεντρωθώ στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία ε, ικανοτήτων στο ψηφιακό τομέα. Ξέρετε ότι έχουμε 17. Λείπουν μάλιστα και τρεις μεγάλες χώρες που δεν υπάρχει τέτοια εθνική συμμαχία. Σε όλες τις χώρες πρέπει να υπάρχει αυτή. Γιατί μόνο με τη συμμαχία αυτή θα μπορέσουμε να φροντίσουμε να εντοπίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές και να ενώσουμε τον κόσμο, κυρίως το ψηφιακό, για να προτείνει δουλειές για τους νέους. Επίσης, έχω ευαισθητοποιηθεί ιδιαίτερα και όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συμπληρωματική ερώτηση. Ναι. Ευχαριστώ. Δεύτερη ερώτηση. Ναι, θέλουμε να προστατεύσουμε επίσης το copyright, τη δημιουργία, τα πραγματικά δικαιώματα, αλλά νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με διάλογο με τις πλατφόρμες. Οπότε πρέπει να υπάρχει και το κατάλληλο θετικό πλαίσιο. Υπάρχει όμως και μια πτυχή. Μέσω του προγράμματος Media πρέπει να στηρίξουμε και την παραγωγή και διανομή. Θα ήθελα να μάθω πώς θα μπορούσαμε μέσω του Media να δώσουμε οικονομική στήριξη και κυρίως να χρησιμοποιήσουμε το νέο χρηματοοικονομικό εργαλείο που μέχρι τώρα επιτρέπει μόνο σε δύο φορείς να συμμετάσχουν στον αντίστοιχο διαγωνισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Γκάμπριλ να απαντήσει. Για να είμαι ειλικρινής, σας σκέφτηκα και αυτή την ερώτηση όταν ε, στις γραπτές μου απαντήσεις ε, συντόμεψα το κομμάτι, γιατί έπρεπε να υπάρχει ένα κομμάτι για τη Δημιουργική Ευρώπη και το Μέντια. Είναι ένα από τα συμβολικά προγράμματα που έχουμε, ακόμη και να έχει μικρό προπολογισμό, 100.000 το χρόνο, η προβολή είναι τεράστια. Και πολλά μένουν να γίνουν. Ναι, το πρόγραμμα Media υπάρχει από το 1991. Πολιτιστική πολυμορφία και πρόθεση των δικών μας ταινιών, του δικού μας πολιτισμικού τομέα. Έχουμε συγκεκριμένο παράδειγμα με το μηχανισμό εγγύησης για την περίοδο 2016-2020. Έχουμε τα μέσα που επιτρέπουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πολιτισμό να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και το έχουν κάνει με εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Θα στηρίξω λοιπόν από φέτος μαζί με το Ταμείο Επενδύσεων και με το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, προκειμένου να υποστηριχτούν τέτοιες πρωτοβουλίες. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Άσλι Φόξ έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Γκάμπριελ, συγχαρητήρια για τον ορισμό σας αυτό. Μπορείτε παρακαλώ να εξηγήσετε στην Επιτροπή μας τις απόψεις σας για τις τεχνολογίες κατανομής. Εσείς πώς βλέπετε τα ωφέλη για τους καταναλωτές. Τι έχετε να πείτε για την απορρίθμιση. Σύντομη ερώτηση, απάντηση τώρα κύριε Γκάμπριελ. Ευχαριστώ κύριε Φόξ για την ερώτησή σας. Αυτό είναι ένα θέμα που με τον Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκης που είναι για τα οικονομικά και τον Αντιπρόεδρο Γιούροβα που είναι για την προστασία του ιδιωτικού βίου έχουμε δουλέψει. Σήμερα ε, μπορούμε με ενθουσιασμό να κοιτάξουμε τις εξελίξεις της τεχνολογία αυτή, από την άλλη μεριά να φροντίσουμε και για την προστασία. Μπορεί να υπάρξει πρόοδος στο τομέα της υγείας, για παράδειγμα, αλλά πρέπει να είμαστε και ειλικρινεί. Είναι ένας κλάδος σε πλήρη εξέλιξη. Με ρωτάτε αν θα ρυθμίσουμε την τεχνολογία. Όχι. Εμείς είμαστε υπέρ της τεχνολογικής ουδετερότητας, όμως παρακολουθούμε από κοντά τις σημερινές εξελίξεις. Και ακριβώς γι' αυτό ασχολήθηκα και έμαθα πολλά. Στην ε, πρώτη διάσκεψη που έλαβε χώρα εδώ, τον Μάιο, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που επιβεβαίωσε τη δέσμευσή μας από αυτού. Έπειτα, θα παρακολουθώ την τεχνολογία αυτή και για να εντοπίσω τι ρυθμίσεις υπάρχουν ήδη, το GDPR για παράδειγμα, όταν μιλάμε για την εμπιστευτικότητα ε, των προσωπικών δεδομένων. Δεν έχει σημασία αν πρόκειται για blockchain ή όχι. Και από την άλλη μεριά πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν και αρνητικές επιπτώσεις από τέτοιες τεχνολογίες. Και εδώ αναφέρομαι σε αυτά που επιτρέπονται, δομή διαφάνεια και εκείνες που δεν επιτρέπονται, το bitcoin, το e-wallet και άλλα που μας υποχρεώνουν να περνάμε από άλλου μέσα, know your customer. Know your customer. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα προσέξουμε και να στηρίξουμε τις θετικές πτυχές από τις οποίες μπορούν να προκύψουν ωφέλη για όλους. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Υπάρχει συμπληρωματική ερώτηση, κύριε Φόξ. Ευχαριστώ. Κυρία Γκάμπριελ, είπατε απαντώντας ότι εγώ ήθελα ρύθμιση. Δεν είπα αυτό. Και να αν συμφωνείτε ε, μαζί μου ότι πολύ συχνά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, κοιτάμε τις νέες τεχνολογίες σαν μια απειλή. Εσείς αναφέρεστε κάπως αρνητικά σε νέες τεχνολογίες. Πολύ συχνά όμως, όταν εμείς οι πολιτικοί αντιστεκόμαστε στον ε, πειρασμό, είναι τότε που βλέπουν το ωφέλη πολίτες. Συμφωνείτε λοιπόν μαζί μου ότι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της FinTech ε, Task Force ήταν να περιμένουμε να δούμε. Θα ήθελα να γίνει το ίδιο και με το DLT, ώστε εμεί οι πολιτικοί να μην καταστρέψουμε κάτι από το οποίο μπορούν πραγματικά να επωφεληθούν οι πολίτες. Ευχαριστούμε πολύ για την, τα σχολεία σας ή οριστής επίτροπος. Εγώ δεν βλέπω τις νέες τεχνολογίες σαν απειλή, αλλά κάθε φορά πρέπει να επανέρχομαι σε αυτό που είπα και στην αρχή, ότι ως Ευρώπη έχουμε ρόλο να παίξουμε οι αρχές μας, οι αξίες μας, η ασφάλειά μας, είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να αμφισβητούνται. Οπότε εγώ προσωπικά πιστεύω πράγματι ότι πρέπει να διατηρήσουμε τον ενθουσιασμό και την αισιοδοξία για να προωθήσουμε τις νέες τεχνολογίες, αλλά αυτό να γίνεται πάντα βάση ανάλυσης η οποία να μας επιτρέπει να μην αποκλείουμε κάποιους από τις αλλαγές αυτές. Αυτή είναι μια αρχή πάνω στην οποία επιμένω πάντα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Επόμενη ερώτηση, Ντίτα Τσαράντζοβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και κύριε Οριστή Επίτροπε. Συγχαρητήρια για τον ορισμό σας πρώτα απ' όλα. Τώρα εσείς ξεκαθαρίζετε ότι αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντική είναι η ψηφιακή ενιαία αγορά για την ευρωπαϊκή οικονομία, την ευρωπαϊκή ανάπτυξη και τις δουλειές στην Ευρώπη. Επίσης είπατε ότι τα δεδομένα πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρώπη. Έχετε δίκιο. Το κέντρο της ανάπτυξης της ψηφιακής αγοράς είναι τα δεδομένα. Αυτά ε, αποτελούν και την ψηφιακή αγορά. Όποτε συμφωνείτε μαζί μας ότι η ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων πρέπει να είναι και δωρεάν στην Ευρώπη. Ρωτά όμως. Επιβεβαιείτε ότι στηρίζετε και συμφωνείτε με τον κύριο Αντσίπ ότι όλα αυτά πρέπει να συνοδεύονται από νομοθετική πρόταση που θα έρθει ακόμα φέτος. Ευχαριστούμε. Απάντηση, η κυρία Γκάμπριελ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Σαράντσοβα. Είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και σήμερα, γνωρίζοντας πώς έχει η κατάσταση, θα ήθελα και να το επιβεβαιώσω. Ναι, είμαστε κατά της ε, τοποθέτησης των δεδομένων της, του εντοπισμού της ε, τοποθεσίας των δεδομένων. Πρόκειται για μια ακόμα ελευθερία. Και για να υποφεληθούμε από την ελευθερία αυτή και να μην υπάρχει γεωγραφικός αποκλεισμός, πρέπει να δούμε ότι υπάρχει. Οπότε δεσμεύομαι ότι από το φθινόπωρο θα πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, θα καθορίσουμε πολύ καλά το που υπάρχει αυτός ο γεωγραφικός αποκλεισμός και θα τον καταπολεμήσουμε. Και υπάρχει και κάτι ακόμα σημαντικό, το δικαίωμα στην μεταφορά του περιεχομένου και η δυνατότητα πρόσβοσης όταν πρόκειται για ρυθμισμένα μέτρα, για παράδειγμα για φορολογικούς λόγους. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί σήμερα μερικές φορές όταν κοιτάμε το θέμα αυτό του γεωγραφικού περιορισμού για τους καταναλωτές, για τις επιχειρήσεις, λένε ότι τους προσφέρει ασφάλεια. Όχι, ο περιορισμός αυτός δεν σημαίνει περισσότερη ασφάλεια. Είναι σημαντικό να το ξέρουμε αυτό, γιατί δημιουργεί φραγμούς εκεί όπου δεν υπάρχουν πια φυσικοί περιορισμοί. Οπότε έχουμε δουλειά να κάνουμε σε αυτό και το λέω, γιατί όταν μιλάμε για το γεωγραφικό αποκλεισμό είναι αυτή η εικόνα της κορυφής του παγόβουνου και ξεχνάμε το τι υπάρχει από κάτω. Όταν κοιτάμε μόνο ότι περισσεύει πάνω από την επιφάνεια του νερού, ξέρουμε 50 πρακτικές που είναι ήδη γνωστές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με περιορισμούς από τις χώρες μέλη, αλλά υπάρχει και ένα μεσαίο κομμάτι όπου επιχειρήσεις επειδή φοβούνται ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος κίνδυνος, νομίζουν ότι πρέπει να κάνουν αυτό τον περιορισμό και στη συνέχεια έχουμε ένα τεράστιο κομμάτι παρακάτω που είναι αόρατο και που έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Υπάρχει συμπληρωματική ερώτηση από την κυρία Σαράντσοβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ για τα ανθερητικά σας λόγια. Όμως αναρωτιέμαι, θα μπορούσατε να είσαστε και πιο συγκεκριμένοι για το τι μέτρα πρέπει να εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να διασφαλίσει ότι η αγορά δεδομένων στην Ευρώπη μπορεί να αυξηθεί. Ευχαριστούμε κύριε Γκαμπρίλ. Όπως το είπα και στην αρχή, τα στοιχεία που έχουμε από την οικονομία δεδομένων είναι 272 δισεκατομμύρια και περιμένουμε πάνω από 640 μέχρι το 2020. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν κάνει τίποτα η Ευρώπη, η αύξηση θα υπάρξει. Άρα καλά θα κάνουμε να επιταχύνουμε. Και γι' αυτό και είπα ότι το πρώτο είναι να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον ε, γεωγραφικό αποκλεισμό που δεν έχει νόημα ύπαρξης. Δεν λέω ότι θα είναι εύκολο. Πρέπει να δουλέψουμε με τις επιχειρήσεις, πρέπει να δουλέψουμε και με τις χώρες μέλη. Κυρία Σαράνσοβα, σα ε, διαβεβαιώ. Υπάρχει ήδη μελέτη αντικτύπου. Έχουμε ήδη κάποιε πρώτε αναλύσει. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, αλλά για μένα δύο είναι σημαντικά τώρα. Ότι για πρώτη φορά σε σχέση με πριν από 1,5 χρόνο όλε οι χώρε συμμετέχουν και το ένα τέταρτο αυτών που απάντησαν είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σήμερα μένει να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο αυτό για να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις. Ευχαριστούμε. Η Ματίνα Μίχελς. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Γκάμπριελ, μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξετάσει τις βασικές αρχές, προστασία δεδομένων, ουδετερότητα δικτύου από την πλευρά της εσωτερικής ενιαίας αγοράς. Δεν είναι όμως κάτι συνολικό. Γιατί υπάρχει και το θέμα της πρόσβασης στον πολιτισμό, στην έρευνα, ε, τα οποία ξεφεύγουν από την αξιολόγηση αυτή. Στο σημείο 7 των απαντήσεών σας λέτε ότι χρειάζεται εξυγχρονισμό των δικαιωμάτων του δημιουργού, ε, μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες, συλλογές κλπ. Δεν υπάρχουν. Σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αρχές αυτές μπορούν να αποθηκεύουν ψηφιακά, αλλά μόνο για λόγους συλλογής και αρχείων. Πιστεύετε ότι η ψηφιακή δυνατότητα σε ένα σύγχρονο κόσμο δεν είναι πολύ περιορισμένη, δεδομένου ότι πρέπει να υπάρχουν πολιτιστικές ανταλλαγές. Ευχαριστούμε. Απάντηση. Ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Και εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το τοπίο έχει αλλάξει. Των πλατφόρμων, των μέσων ενημέρωσης, των υπηρεσιών, δικαιώματα δημιουργών. Πώς να βρούμε σωστή ισορροπία για όλους, για να μπορούν όλοι να συμμετέχουν σε αυτή την ψηφιακή αλλαγή. Θέτεται και ένα ζήτημα πάνω στο οποίο θέλω να συνεχίσω να δουλεύω και περισσότερο μάλιστα ακόμα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, με τους ενδιαφερόμενους. Πραγματικά θέλω να ακούσω όλες τις πλευρές και δεσμεύομαι γι' αυτό. Αν επιβεβαιωθεί ο ορισμός μου, θέλω όλοι όσοι έχουν ακόμα πράγματα να πούν, να τα πούν, να μπορέσουν να εκφραστούν. Γιατί πιστεύω ότι κι εσείς το δείξατε ακριβώς με αυτά που είπατε. Υπάρχουν πτυχές σχετικά με τις οποίες δεν έχουμε δώσει αρκετές, ε, αρκετή προσοχή, άλλες που παραμένουν κρυφές. Γι' αυτό εγώ θέλω τη συμμετοχή όλων. Είναι ένα βασικό θέμα για μένα. Είναι ένα από τα θέματα πάνω στον οποίο το λέω ότι θέλω να συνεχίσω να δουλεύω για να καταλάβω καλά τι παίζεται πλήρως. Η αρχή πάντως υπάρχει. Πρέπει να βοηθήσουμε τους δημιουργούς για καινοτομία και για δημιουργία. Να ανταμείβονται σωστά για το έργο τους και τη δημιουργία τους. Να επιτρέψουμε την έρευνα στις βιβλιοθήκες, σε ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς που συμμετέχουν στην ταυτότητά μας και στην αριστεία μας. Πρέπει να συνεχίσουν να μπορούν να το κάνουν. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής για αυτά τα ζητήματα. Θέλω να δουλέψω περισσότερο πάνω σε αυτά για να ακούσω και τους υπόλοιπους, να ακούσω όλες τις απόψεις. Ήταν πολύ χρήσιμο τις τελευταίες εβδομάδες και θα συνεχίσω προς την ίδια κατεύθυνση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει συμπληρωματική ερώτηση, κυρία Μίχελς. Να μένω με ενδιαφέρον αυτή τη συνεργασία. Αναφερθήκατε στην ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της κοινή γνώμης και στον ε, τομέα των πολιτισμικών αγαθών ε, αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο ε, πρόβλημα με το Euronews και την εξαγορά του BBC όπου υπάρχουν δηλαδή επιπτώσεις ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού αλλά και την επιτελμορφία των προγραμμάτων. Εσείς λοιπόν θα αναλάβετε δράση σε αυτό το τομέα. Η κυρία Γκάμπριλ, ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή κυρία Μίχελς είναι πολύ σημαντική και ευαίσθητη. Σημαντική γιατί το γνωρίζουμε ότι έχει αποστολή το Euronews και είναι ευρωπαϊκό αυτό, γιατί προτείνει ε, πληροφορίες και ενημέρωση ποιότητας. 38% των Ευρωπαίων θεωρούν ότι ενημερώνονται ικανοποιητικά και το νούμερο αυτό πρέπει να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Υπάρχει συμφωνία σήμερα με το Euronews που υπογράφηκε το Φεβρουάριο του 2017 για τις τέσσερις επόμενες χρονιές. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε εντοπίσει στόχους και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρεί το Euronews και ήταν έξι και πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να παρέμβει ανα πάσα στιγμή. Για μένα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φροντίσουμε να τηρείται αρχή της πολυγλωσσίας, ε, να προστατεύονται δημοσιογράφοι, να μην υπάρχουν απολύσεις. Κάποια στιγμή ακούσαμε ότι υπήρχαν. Πρέπει επίσης να φροντίσουμε η αποστολή του Euronews που ε, διακόπτει η Πρόεδρος. Α, συγγνώμη, κυρία Γκάμπρελ, ξεπέρασα το χρόνο μου. Ναι, απλώς επιβεβαιώνω ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που θέλω να κάνω εφόσον όριστο είναι να συζητήσω περισσότερο το θέμα αυτό του Euronews. Γιατί πρέπει μαζί σας να διασφαλίσουμε την συνέχεια του Euronews στην αποστολή του. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο σε ένα λεπτό να απαντήσει κανείς σε τέτοια θέματα. Λυπάμαι που χρειάστηκε να σας περιορίσω. Συνεχίζουμε λοιπόν. Η κυρία Τζούλια Ρέντα τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Οριστής Επίτροπο, έχω καταλάβει ότι λέτε κι εσείς πως χρόνια μόνο μένουν για την αποστολή σας, δύσκολα θα ολοκληρώσετε όλα όσα μένουν να ολοκληρωθούν. Αλλά υπάρχουν και κάποια δύσκολα ζητήματα ε, που όμως απασχολούν το κοινό. Τα ε, δικαιώματα στην ε, προστασία των δεδομένων, το θέμα της κρυπτογράφησης. Ακούγονται μερικά αντιφατικά. Ρώτησα και συνάδελφοι το ε, ο άρθρο 13 ε, του copyright ευθυγραμμίζεται με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλοι συμφωνούν ότι οι δημιουργοί πρέπει να πληρώνονται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ελέγχονται και όλα όσα μπαίνουν online. Είναι πολύ σημαντικό το περιεχόμενο για τους πολίτες και για την καινοτομία. Τι θα κάνετε λοιπόν, θα παρεύετε στις χώρες μέλη και θα προτείνετε νομοθεσία όπως έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία στην εφαρμογή σε όλες τις χώρες μέλη. Ευχαριστούμε, κυρία Γκάμπριελ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ρεντά, για την ερώτησή σας. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και ελπίζω όντω να υπάρχουν ακόμα σημεία ε, στο οποίο δεν θα αποφασίζουμε από πάνω προς τα κάτω, η συζήτηση πρέπει να συνεχιστεί. Και γι' αυτό φτάνω, μένω ακόμα δύο χρόνια στη θητεία της Επιτροπής αυτής, έχω σχηματίσει κάποια γνώμη από τις επαφές μου μαζί σας και με τους εμπειρογνώμονες στην Κομισιόν. Δεσμεύομαι για διάλογο και νομίζω ότι το δείχνω ότι σκοπεύω να πάω προς αυτήν την κατεύθυνση. Τώρα για το e-commerce, την οδηγία αυτή για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Καταλαβαίνω πόσο μεγάλη σημασία έχει για την ψηφιακή ενιαία αγορά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Είναι το νομικό πλαίσιο που επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία μέσα στην αγορά αυτή. Το ζήτημα που τίθεται σήμερα είναι θα αναθεωρήσουμε την οδηγία ή όχι. Η απάντηση έχει δοθεί. Γιατί ήδη έγιναν τρεις αξιολογίες το 2010, το 2012 και το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ότι είναι κατάλληλη ακόμα η οδηγία. Εξάλλου το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο από τη δικιά του την πλευρά την υποστήριξαν αυτή την οδηγία. Σήμερα είμαστε αντιμέτωποι με νέα πραγματικότητα και γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει συνοχή. Αναφέρθηκα και στην περιορισμένη ευθύνη των πλατφορμών και την αφαίρεση του παράνομου περιεχομένου. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα αυτό σήμερα. Είναι σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μπορούμε να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά τι μπορούν να κάνουν οι χώρες μέλη. Αντιλαμβάνομαι ποιε είναι οι αξίες μας, δεν θέλουμε γενική εποπτεία, η οδηγία είναι σε αυτό. Αλλά πρέπει να παρακολουθούμε όμως το τι γίνεται στις χώρες μέλη θα αντιδράσω στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου. Και θα αντιδράσω όταν βλέπω ότι σε θέματα που είναι αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν τηρούνται οι κανόνες. Διακόπτει η Πρόεδρος. Λυπάμαι, πρέπει να σας διακόψω, κυρία Γκάμπριελ. Υπάρχει συμπληρωματική ερώτηση. Ε, είμαι περίεργη όμως κατά πόσο θα υπάρξει τελικά νομοθεσία για την αφαίρεση περιεχομένου αλλά θέλω και ένα δεύτερο, γιατί είμαι από δύο επιτροπές βλέπετε σήμερα, η ασφάλεια στο κυβερνοχώρο. Στις γραπτές απαντήσεις απαντήσατε για την ασφάλεια αυτή και ρωτάω, θα κάνετε προτάσεις για να βελτιώσετε την ε, ασφάλεια στο διαδίκτυο. Η ευθύνη Επίσης εκείνων που δεν φροντίζουν να αντιμετωπίσουν τα θέματα της ασφάλειας ε, στο διαδίκτυο σε ό,τι τους αφορά στις δικές τους δηλαδή αρμοδιότητες. Απάντηση. Ευχαριστώ, είναι μια δύσκολη ερώτηση. Ναι, θα υπάρχει αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής το Σεπτέμβριο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Μπορώ να επανέλθω στην εντολή της ΕΝΗΣΑ, στην πιστοποίηση και τη σήμανση αλλά το συνδέσατε αυτό και με την ευθύνη των προϊόντων. Οπότε, έτσι επανέρχεστε σε θέματα για το οποίο χρειάζεται ε, ε, ε και άλλη συζήτηση. Όταν ένα αυτοκίνητο συνδεδεμένο περνάει τα σύνορα, τα δεδομένα μεταφέρονται. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να συνεχίσει η συζήτηση σε αυτό. Λοιπόν, εγώ το είπα, στα πλαίσια της ε, αναθεώρησης που θα προτείνω, θα υπάρξει αυτή η πιστοποίηση, αυτή η σήμανση, θα υπάρχει η αναθεώρηση της εντολής της ΕΝΗΣΑ και θα προτείνω ενίσχυση του πλαισίου των ε, εθνικών κέντρων σε περίπτωση ατυχήματο. Έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και στη συνέχεια Όσον αφορά την ευθύνη για τα προϊόντα, ας μιλήσουμε με όλους τους ενδιαφερόμενους για να μην τους επιβάλλουμε μία λύση που δεν θα είναι κατάλληλη και που δεν θα λαμβάνει υπόψη τα δικά τους συμφέροντα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και πάλι ο λόγος στον ε, Μάρκο Τσούλο τώρα. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, έχουμε τριμερή διάλογο για το κανονισμό για το geo-blocking, για το γραφικό εντοπισμό, ιδιαίτερα στο τηλεοπτικό περιεχόμενο βάση εθνικού περιεχομένου, όταν έχουν σύμβαση αυτή η πάροχη περιεχομένου με τρίτους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τώρα έχει αναλάβει, μάλλον έχει θετήσει αποφάσεις αναπερίπτωση, χωρίς μια συνολική οργα... Ε, προσέγγιση συγγνώμη, για το θέμα. Χωρίς να εξετασάδει σε βάθος τις υποθέσεις αυτές και τις ρήτρε γεωγραφικού εντοπισμού. Δεν θέλω τώρα να αναφερθώ συγκεκριμένα στο επιχειρηματικό μοντέλο, αλλά θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να ξέρουμε εάν και πότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει ξεκάθαρη και σαφή απόφαση σε σχέση με αυτέ τι ρήτρε που αφορούν το geo το γεωγραφικό εντοπισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Γκάπριλ για την απάντηση. Κύριε Τζούλο, ευχαριστώ. Θα χωρίσω την ερώτηση αυτή σε δύο τμήματα. Καταρχάς, να μιλήσω για την έκθεση για το geo-blocking και να επενθυμίσω το στόχο αυτού του κανονισμού. Στόχος είναι η προστασία των δικαιωμάτων των εμπορευομένων και των καταναλωτών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, συγκεκριμένες υποθέσεις που αφορούν ακριβώς την παθητική πώληση προϊόντων. Αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι να έχουμε σαφήνεια, το είπε και η Κομισιόν, ότι από τη στιγμή που υπάρχουν κίνδυνοι παράκαμψης, οποιαδήποτε συμφωνία συνάπτεται μεταξύ παραγωγού και διανομία ακυρώνεται. Άλλο τώρα να μιλάμε για τα απτικοακουστικά. Δεν έχουμε ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν μια διάκριση, ένα διαχωρισμό. Πρέπει λοιπόν να ε, υπενθυμίζουμε ότι εμείς μελετήσαμε συγκεκριμένες υποθέσεις, συγκεκριμένε περιπτώσεις, η Γενική Διεύθυνση για τον Ανταγωνισμό έκανε τη δουλειά της και δεν εφαρμόσαμε μέτρα γενικού χαρακτήρα, αλλά η κάθε περίπτωση εξετάστηκε μεμονωμένα. Οπότε θα πρέπει να διακρίνουμε, πιστεύω, τις να ξεχωρίσουμε τις παθητικές πωλήσει από τα οπτικοακουστικά όσον αφορά την αρχή της διαφύλαξης των γεωγραφικών αδειών και τα οπτικοακουστικά. Πάντως εγώ είμαι έτοιμη για κάθε υπόθεση της οποίας λαμβάνω γνώση να το συζητήσω και με τους άλλους συναδέλφους επιτρόπους και ιδιαίτερα με την κυρία Βεσταγκέρ. Ευχαριστώ. Με δευτερολογία του κυρίου Τσούλο. Ναι. Να κάνω πιο άμεση την ερώτησή μου. Ρωτάω στο μέλλον Αναμένουμε μια νομοθετική πρόταση από την Κομισιόν, η οποία θα επιτρέπει ακριβώ την υπέρβαση των γεωγραφικών αδειών στα οπτικοακουστικά. Είναι έτσι. Η κυρία Γκάμπριελ, απαντήστε παρακαλώ. Κοιτάξτε ειλικρινά, από τι ξέρω σήμερα και βασιζόμενοι στις συζητήσεις που είχα και με τους εμπειρογνώμονες αλλά και με τους διάφορους ειδικού, αυτό δεν προβλέπεται για το άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ. Το επόμενο πεντάλεπτο από τον Σάνθο Γιάννου Σκόρμιν Μικέ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ θα πρέπει να αντιληφθούμε πόσο πίσω βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Και ποιος είναι ο λόγος γιατί στις Ηνωμένε Πολιτείες κανένας δεν ασχολούνταν με την ισότιμη πρόσβαση. Όποιος ήθελε δηλαδή πήγαινε και αγόρασε το δικό του σύστημα από μια ιδιωτική επιχείρηση και έτσι ε, έχει καταφέρει αυτή η χώρα να είναι πιο ανεπτυγμένη σε ό,τι αφορά αυτές τις ε, πολιτιστικές υπηρεσίες σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα μας λέτε από την άλλη πλευρά ότι θα πρέπει οι συγγραφές να λαμβάνουν ε, την κατάλληλη αμοιβή. Ποιος θα καθορίζει το επίπεδο αυτής της κατάλληλης αμοιβή. Από εκεί και μετά αναφερθήκατε στη ρητορική μίσους. Ε, ποιος και πάλι θα ορίσει την ρητορική ε, μίσους ως τέτοια. Ε, ρητορική μίσους είναι για παράδειγμα να πούμε ότι οι Εβραίοι προσπαθούν να ελέγξουν ε, τον παγκόσμιο τραπεζικό τομέα ή όταν λέμε ότι θέλουμε να επιβάλλουμε υψηλή φορολογία στις διεθνείς επιχειρήσεις. Είναι ρητορική μίσους όταν όταν λέμε ότι η Ρωσία προσπαθεί να εισβάλλει στην Ευρώπη. Ποιο λοιπόν θα είναι εκείνο που θα κληθεί να ορίσει το τι είναι ρητορική μίσου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο, κυρία Γκάμπριελ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση αυτή. Θεωρώ ότι στην κοινωνία μας, στην δημοκρατική, δεν έχει θέση το μίσος. Εμείς διευρύνουμε ακριβώς τον ορισμό ώστε εκεί να περιλαμβάνονται οποιοσδήποτε παραπομπές, ε, εθνοτική προέλευση, σεξουαλικότητα, οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να προσβάλλει κάποιον. Αυτές οι ομιλίες μίσους νομίζω ότι προσβάλλουν ακριβώς την βάση της δημοκρατικής μας κοινωνίας. Να βεβαίως η ελευθερία έκφρασης πρέπει να προστατεύεται, η ελευθερία ενημέρωσης. Επίσης, ταυτόχρονα όμως, για τις ομιλίες μίσους θα πρέπει να είμαι ξεκάθαρη ότι θεωρώ ότι εδώ ακριβώς θα πρέπει να προασπίσουμε όλοι μας το δικό μας το πρότυπο, της κοινωνίας μας, τις αξίες μας και τις αρχές μας. Θα σταματήσω εδώ πραγματικά γιατί νομίζω ότι ο σεβασμός ε, του άλλου όταν έχετε κάτι να πείτε πρέπει να αποφεύγει οποιαδήποτε ομιλία μίσους. Αυτό είναι κάτι για το οποίο δεσμεύομαι να εργαστώ περισσότερο. Τώρα, για τις επιπτώσεις αυτών των ομιλιών μίσους στα παιδιά, για τις επιπτώσεις ακριβώς που έχουν σήμερα αυτές οι ομιλήσεις, οι ομιλίες μίσους σε ανθρώπους που έχουν το μέλλον μπροστά τους. Θα ήθελα εδώ να κάνω έκκληση στην ευθύνη όλων μας, γιατί πραγματικά πρόκειται για ένα θέμα με το οποίο δεν γίνεται να παίζουμε απλά και μόνο. Ευχαριστώ κύριε και θέλετε να δευτερολογήσετε. Ναι, δυστυχώς δεν έλαβα μια συγκεκριμένη απάντηση. Είμαι πολύ μεγαλύτερη ηλικία από εσάς, ε, κυρία Και βρέθηκα ε, στη φυλακή ε, κατά την περίοδο του κομμουνισμού και ένας από τους, μια από τις κατηγορίες που μου απαγγέλθηκαν ήταν ότι είχα διαβάσει πληροφορίες οι οποίες θεωρούνταν πολύ σημαντικές για την ασφάλεια της δικής μου χώρας. Και μου επιβλήθηκε πρόστιμο 9.000 ευρώ με το γεγονό ότι διέθεσα πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες σε δημοσίω σε ό,τι αφορά ε, την, ε, το επίπεδο νοημοσύνης, το δίκτυο νοημοσύνης ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οπότε αυτό που ρωτώ και ξαναρωτώ είναι ποιος θα αποφασίζει ως προς το τι είναι ψευδής είδηση ή ψευδής πληροφορία και ε, ποια πληροφορία δεν είναι ψευδής ή ποια πληροφορία τελικά είναι σημαντική για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι τελικά δεν θα πρέπει ο καθένα να μπορεί να πει αυτό που θέλει και από εκεί και μετά να λαμβάνει την ευθύνη για τα όσα λέει. Κυρία δεν έχει το λόγο. Είμαι υπερήφανη, υπερήφανη που προσπίζομαι την, ε, τις αρχές ισότητας μεταξύ άντρων και γυναικών. Και όπως είπα... Όπως είπα σήμερα, δεν πρέπει να πούμε ποιος είναι υπεύθυνο και ποιος όχι. Αυτά που ανέφερα εδώ είναι αρχές αυτορύθμισης και αυτό είναι δική μας ευθύνη. Ναι, πράγματι έχουμε αξίες που θα πρέπει να πρασπιστούμε και εγώ θα πρασπιστώ τις αξίες μέχρι τέλους. Σας ευχαριστούμε θερμά. Αντώια Σουάπτουρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, κυρία Αριστήσα ε, Επιτρόπε, εγώ δεν θα θέσω ένα ερώτημα το οποίο θα οδηγήσει σε απάντηση με χειροκροτήματα. Ε, ε μετά από τα 8 χρόνια τα οποία σας γνωρίσαμε από την πλευρά ε, του ΕΛΚ ε, θεωρούμε πως ε, τα δύο χρόνια που θα έχετε στη διάθεσή σας ως Επίτροπος θα είναι υπεραρκετά για να επιτύχετε κάποια πράγματα. Η ενδιάμεση αναθεώρηση από την πλευρά της Επιτροπής έθεσε και κάποια ερωτήματα. ερωτήματα στα, σε σχέση με τα οποία έχετε λάβει τώρα από τον προκάτοχό σας τον κύριο Έτιγκερ έξι νομοθετικέ προτάσει οι οποίε τρέχουν και για τι οποίε αναμένουμε κάτι από εσά. Ακριβώ λοιπόν σε σχέση με αυτή την ενδιάμεση αναθεώρηση θα ήθελα να σα ρωτήσω τι ε, θέλετε να κάνετε ω επίτροπο σε σχέση με αυτό το, ε, την platform του business και την platform του consumer ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις αθέμητε εμπορικές πρακτικές. Και επίση, μπορείτε να μα επιβεβαιώσετε ότι θα δώσετε περαιτέρω συνέχεια στην ενδιάμεση αναθεώρηση τη Επιτροπή σε σχέση με την πλατφόρμα αλλά και το e-sector inquiry. Ευχαριστούμε. Ε, κυρία Γκάμπρελ, έχει το λόγο για να απαντήσει. Κύριε Σφαμπ, ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, αυτό είναι μήμα της ταυτότητάς μου η εμπειρία στο ΕΛΚΑ, αλλά επίσης είναι εξίσου και η θαυμάσια συνεργασία που είχαμε τους συναδελφούς των υπολείπων πολιτικών ομάδων και αυτό τελικά μας χαρακτηρίζει όλους. Το να δούμε δηλαδή ακριβώς το πώς θα προσπιστούμε τα συμφέροντα στις διάφορες πολιτικές των πολιτών. Και σήμερα είχα την ευκαιρία να απαντήσω, αλλά θέλω να επανέλθω ακριβώς για να κάνω και διευκρινήσεις ότι θα υπάρξει πρόταση Κομισιόν σε σχέση με αυτές τις θέμητες πρακτικές που αφορούν τις πλατφόρμες και τις επιχειρήσεις. Είναι λοιπόν εξίσου σημαντικό να προασπίσουμε και τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των ε, καταναλωτών. Αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Και θα το πω αυτό με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Όταν επιλέγουμε ένα ξενοδοχείο, θα έπρεπε να γνωρίζουμε αν η προσφορά η οποία μας υποβάλλεται ανταποκρίνεται πραγματικά στα δικά μας τα κριτήρια ή αν μα δίνουν αυτή την προσφορά επειδή ήταν οι πιο διαφημισμένοι. Αυτή είναι η διαφορά. Επειδή θεωρώ ότι αυτό ακριβώς είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να, να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή καταναλωτής, επιχείρηση, επειδή ακριβώς, εδώ ακριβώς θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, θα πρέπει να υπάρχουν οι συνθήκες που θα επιτρέπουν την καινοτομία και την δημιουργία. Θα προσπιστώ λοιπόν αυτές τις αρχές και χρειάστηκε να περιμένω λίγο στην μετάφραση την ερώτησή σας για την πληροφορική. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα αντιμετωπίσω συλλογικά και με άλλους επιτρόπους, ακριβώς ώστε να διατηρήσουμε τις πλατφόρμες ως δημιουργούς και καινοτόμους ποικίλου περιεχομένου, αλλά ταυτόχρονα δεν θα διστάζουμε να λαμβάνουμε μέτρα και αποφάσεις όταν υπάρχουν προβλήματα, είτε περιορίζοντας τις δραστηριότητε, είτε βοηθώντας τους καταναλωτές. Ε, θέλετε να δευτερολογήσετε κύριε Ράσφα. Ναι. Ε, σε ό,τι αφορά την απάντηση που δώσατε σε ό,τι αφορά το ρόλο της πλατφόρμας ως Gatekeeper θα υπάρχει, θα συγκαταλέγεται εκεί και ένας έλεγχος ε, του αλγορίθμου. Ε, δεν έχω μία δεν έχω κατασταλάξει σε ό,τι αφορά τη στάση μου, αλλά εγώ θα ήθελα να ρωτήσω εσά ποια είναι η θέση σα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των αλγορίθμων. Η κυρία Γκάμπριλα έχει το λόγο για να απαντήσει. Ευχαριστώ και πάλι για αυτή την ερώτηση. Εγώ δεν το βλέπω μόνο από τη σκοπιά του ελέγχου, αλλά από τη σκοπιά της καλύτερης κατανόησης της λειτουργίας των αλγορίθμων. Και ευχαριστώ το Κοινοβούλιο που μας βοηθάει να το κάνουμε αυτό. Γιατί υπάρχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για τους 16 επόμενους μήνες. Έχουμε μια χρηματοδότηση χάρη ακριβώς στο Κοινοβούλιο για να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς λειτουργούν αυτοί οι αλγόριθμοι που δεν θα πρέπει να αποτελούν το αόρατο χέρι με τις αρνητικές επιπτώσεις που ξέρουμε όλοι. Θα πρέπει να αποτελούν μια απόδειξη αυτών των αξιών ισότητας και διαφάνειας ώστε η προστιθέμενη αξία του ανθρωπίνου όντως της δημιουργική Ευρώπης αφορά ακριβώς τις προσπάθειες που καταβάλουμε. Ευχαριστούμε. Επόμενη τώρα ερώτηση από την Μπέκη Τσίπελ. Σας ευχαριστώ κυρία Γκάμπριελ. Επιτυχή σε μια ψηφιακή αγορά θα πρέπει ταυτόχρονα να διασφαλίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα των ε, πολιτών, ε, στου οποίου απευθύνεται δηλαδή η ελευθερία τη έκφραση, ε, προστασία τη ιδιωτικότητα και των προσωπικών δεδομένων και εμπιστευτικότητα των επικοινωνιών. Πώ λοιπόν εσεί θα διασφαλίσετε συγκεκριμένα την την προστασία των λόγων δικαιωμάτων και συμφωνείτε μαζί μου ότι είναι πραγματικά ζωτική σημασία να προστατευτούν τα δικαιώματα αυτά που επιθετικέ επιχειρήσει όταν θα είναι νέε πρωτοβουλίε στο πλαίσιο τη ενιαία ψηφιακή αγορά και πιο συγκεκριμένα. Ε, τι ακριβώ σχεδιάζετε να κάνετε σε ό,τι αφορά τι δεσμεύσει που αναλάβατε, έτσι ώστε ο κανονισμό για το e-privacy να ε, παρέχει το ίδιο υψηλό επίπεδο προστασία ε, δεδομένων όπως αυτό που έχει διασφαλιστεί για τα προσωπικά δεδομένα, ειδικότερα απέναντι σε λόμπι τα οποία προσπαθούν να υπονομεύσουν διατάξεις οι οποίες ακριβώς έχουν ε, ε, προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα. Με άλλα λόγια, πώς θα προστατεύσετε αυτά τα δεδομένα από τις πρακτικές ε, των λόμπι που προσπαθούν να καταστατηγήσουν κάποια, κάποιες από τις υφιστάμενες διατάξεις που προστατεύουν τα δικαιώματα των πολιτών. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Κυρία Γκάμπρελ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και την ερώτηση. Όπως είπα στην αρχή, για μένα είναι ένα θέμα συνέπειας. Έχουμε το DGPR που θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μάη 18. Εμείς εδώ έχουμε καθορίσει κριτήρια ισχυρά και αφετέρου για λόγους συνάφειας θα υποβάλουμε τον κανονισμό e-privacy που αφορά ακριβώς την εμπιστευτικότητα των επικοινωνιών. Κάτι το οποίο για μένα εδώ είναι κεντρική σημασία είναι η σύμφωνη γνώμη, η συγκατάθεση. Εξάλλου θα δείτε ότι στο e-privacy, το, e το, στο EGDPR, η, συγκατάβαση, η συγκατάθεση έχει τεράστια σημασία. Όταν λέω κάτι τέτοιο, το λέω επειδή ακριβώς είχαμε παλαιότερους ορισμούς του e-privacy που θεωρούμε παροχημένους με αντίστοιχες κυρώσεις κλπ. Οπότε, αν δεν καταλήξουμε σε αυτή την συνέπεια στην οποία αναφερόμουν, τι θα γίνει. Στο DCPR έχουμε εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων που ακριβώς εποπτεύουν την ε, εφαρμογή. Αν το e-privacy δεν υιοθετηθεί, τότε θα έχουμε άλλες αρχές οι οποίες θα το πράξουν, θα πρέπει να πράξουν ό,τι χρειάζεται, γιατί δεν θα μπορέσουν να επαναφέρουν τον, αυτό που κάναμε στο GDPR. Γι' αυτό εγώ το λόγο δεσμεύομαι να συνεργαστώ με το Κοινοβούλιο, ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τα υπολοιπόμενα, τι μένει ακόμα να γίνει να δούμε μήπως αν μας πει κανείς ότι δεν γίνεται, πολύ φιλόδοξο κτλ. Να πούμε ότι κοιτάξτε εδώ έχουμε να κάνουμε την ασφάλεια των πολιτών. Για το οποίο θεωρούν αυτή ως την πρώτη προτεραιότητα της Ευρώπης. Ευχαριστούμε. Κυρία Ζίπελ, δεύτερο ερώτημα. Ναι, σας ευχαριστούμε. Ε, πολύ στο e-privacy αλλά ελπίζω να σα κατάλαβα σωστά σε αυτό που είπατε, ότι δηλαδή εν γέννη θα κάνετε ό,τι μπορείτε προκειμένου να ε, προστατεύσετε την ιδιωτικότητα του πρόεδρου σε όλου του τομείς τη νέας ψηφιακή ε, αγοράς. Επειδή τώρα το και σας είναι πολύ ευρώ, θα ήθελα να σα ρωτήσω ένα ζήτημα που αφορά ειδικότερα την Επιτροπή Γιούρη. Γνωρίζετε πω υπάρχει, ε, έχει ασκηθεί κριτική στον κανονισμό ΚΑΠΣΑΤ, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την αρχή τη χώρα προέλευση, αλλά και σε με άλλα ζητήματα. Εσεί υποστηρίζετε αυτή την αρχή τη χώρα. Ε, ε, και αν ε, ναι, πώ θα αντιμετωπίσετε τι επικρίσει προκειμένου τελικά να δοθεί συνέχεια σε αυτή την πρωτοβουλία και πώ θεωρείτε πω θα συνεχίσει να ισχύει ο κανονισμό στο πλαίσιο και τη της υπόθεσης για το Sky Competition και από εκεί και μετά θεωρείτε ότι ο γεωγραφικός αποκλεισμός και οι σχετικές ρυθμίσεις θα είναι αδύνατες στο πλαίσιο του Sky Competition. Δύσκολη ερώτηση. Καταρχά, λέει κάποιο, θα έχουμε πραγματικά την αρχή τη χώρα προέλευση. Θα πρέπει όμω να διευκρινίσουμε ότι αυτό που προτείνουμε είναι να διευκολύνουμε την λήψη δικαιωμάτων όταν έχουμε να κάνουμε με, διάζοντα, με υπηρεσίες. Δηλαδή το replay και οι υπηρεσίε online. Όπω λέμε ακόμα και στα γαλλικά. Οπότε δεν αφισβητούμε σήμερα την αρχή της χώρας προέλευσης, επειδή ακριβώς θέλουμε να προχωρήσουμε όσον αφορά την κυκλοφορία και τη διανομή, την διασυνοριακή. Ταυτόχρονα όμως γνωρίζω ότι υπήρξαν ανησυχίε που εκφράστηκαν. Μάλιστα πριν μια εβδομάδα ο εισηγητής δεν κατάφερε να καταλήξει συνάντηση. Αυτή η φορά θα γίνει όμω, οπότε είναι σημαντικό να προχωρήσουμε. Αλλά ταυτόχρονα να απαληθεύουμε ακριβώ που είναι τα όρια με το geo-blocking. Σας είπα ότι η αρχή της χώρας προέλευσης δεν σημαίνει ότι περιορίζουμε τη δυνατότητα των συμβάσεων για να περιορίσουμε ακριβώ τη δυνατότητα παρχή περιεχομένου σε κάποιε περιοχέ. Το geo δεν αποτελεί παθητικές πωλήσει. Μιλάμε για πέντε συγκεκριμένες υποθέσεις που θέλουμε να ρυθμίσουμε και θα συνεχίσουμε από αυτού, ώστε κάποιες βασικές ε, αρχές να διασφαλίζονται. Θα πρέπει όμως οπωσδήποτε να προχωρήσουμε εδώ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Επόμενη ερώτηση από Άντζελ Τζαμπάσκη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γκάμπριελ, θα ήθελα καταρχήν να σας συγχαρώ με το γνώσιο ότι έχετε οριστεί ως Ευρωτική Επίτροπος και βέβαια ε, το χαρτοφυλάκιο που έχετε αναλάβει ε, είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά και την ποικιλομορφία. Ένα ζήτημα, δηλαδή ένα χώρο ο οποίο με απασχολεί στο πλαίσιο τη Επιτροπή Πολιτισμού. Ε, τώρα, ε, σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση, χρειαζόμαστε ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, των δημόσιων συστημάτων υγεία στα κράτη-μέλη και αν ναι, τι θα κάνουμε ούτω ώστε να επιταχύνουμε αυτή την ψηφιοποίηση στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Λόγω στην κυρία για να απαντήσει два изключително важни аспекта. Σας ευχαριστώ κύριε Ζαμπάσκη. Πράγματι πολύ σημαντικές ε, αυτές οι τυχές της εννέας ψηφιακής αγοράς. Η αγορά αυτή προφανώς θα πρέπει να έχει ωφέλη για τους καταναλωτές μας. Ε. Ε, και ακριβώ αυτά τα ωφέλη θα αποτελέσουν τις προτεραιότητε ε, για τη δική μου θητεία στου ε, μήνε που θα ακολουθήσουν. Σε ό,τι αφορά το χώρο της υγείας, Προφανώ. εδώ όλοι θεωρούν πως είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα. Όταν κάνουμε δηλαδή λόγο για ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων, τότε θα πρέπει να έχουμε και το θάρρο να κάνουμε ένα βήμα πιο πέρα και να επιτρέψουμε την πρόσβαση στα ε, δεδομένα υγείας ηλεκτρονικά, για παράδειγμα μέσω ε, της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Με αυτόν τον τρόπο, ανάλογα δηλαδή με την κάθε χώρα, ανάλογα με το κάθε νοσοκομείο, ανάλογα με την κάθε κλινική, να αποφύγουμε ε, να, την ανάγκη του να επισκέφτεται ο ασθενής επανειλημμένα το συγκεκριμένο σημείο ή να ε, γίνονται ξανά και ξανά οι ίδιες εργασίες. Από ό,τι γνωρίζω, αυτή αποτελεί και μία από τις προτεραιότητες της Εστονικής ε, Προεδρίας, αλλά είμαι πεπισμένο ότι θα αποτελέσει και μία από τις προτεραιότητε της Βουλγαρικής Προεδρίας. Από εκεί και μετά ε, ο στόχος είναι ε, ούτως ή να εφαρμοστεί και στη Βουλγαρία το, η συλλογιστική του e-health. Οπότε λοιπόν ε, ο τομέας ε, της, του δημοσίου, της δημόσιας υγείας είναι πάρα πολύ σημαντικός ακριβώς για να επιτύχουμε τον στόχο του να υπάρχει ένα σημείο εξυπηρέτησης, να υπάρχει ένας τρόπος Δηλαδή το να έχει κανείς ένα έγγραφο το οποίο το αποστέλει μία φορά και από εκεί και μετά το έγγραφο αυτό διαβιβάζεται μεταξύ των διαφορών υπηρεσιών χωρίς να χρειάζεται ο ενδιαφερόμενος να το αποστέλει επανειλημμένα. Με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης θα εξοικονομεί χρόνο ε, και όταν θα είναι συνδεδεμένος δεν θα ε, σπαταλά ε, πλέον τον χρόνο του. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με το άρθρο 12. Το άρθρο 12 το οποίο θα μας επιτρέψει ακριβώς να μειώσουμε το διοικητικό άρθρο για τους πολίτες μας και να καταστήσουμε πιο αποτελεσματική την ε, εξυπηρέτηση από τις δημοσίες υπηρεσίες. Ε, πιο αποτελεσματική, πιο ακριβή και ε, θα αυξήσουν και την νομιμότητα αυτών των υπηρεσιών απέναντι στους πολίτες. Ευχαριστούμε. Λέει πρόεδρος, επακολουθώ ερώτημα. Τον κύριο Τζαβάσκη. Ναι, σας ευχαριστώ για αυτήν την περιεκτική απάντηση. Ένα συμπληρωματικό ερώτημα. Τι θα κάνει η Επιτροπή προκειμένου να μειώσει το διοικητικό άχθος για τους πολίτες αλλά και τις επιχειρήσεις σε σχέση με τις διασυνοριακές συνάδελφες. Ναι. Ουσιαστικά, απαντώντας σε αυτό το ερώτημα, θα βασιστώ στις απαντήσεις που έδωσα ε, προηγουμένω, Όταν κάνουμε λόγο για διασυνοριακέ ή υπηρεσίε, υπηρεσίες, ε, ουσιαστικά αναφερόμαστε στην Ευρώπη εκείνη που θέλουμε να επιτύχουμε. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη, ε, μια Ευρώπη η οποία εξασφαλίζει πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες για τους πολίτε. Και γι' αυτό εστιάζουμε σε μια σειρά αποζητήματα. Καταρχήν, εφαρμογή τη αρχή που μόλι σα περιέγραψα, δηλαδή μία και μόνη αποστολή ενό εγγράφου, άπαξε και διαβατω Με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης δεν ναι, χρειάζεται να επαναλαμβάνει τις ίδιες εργασίες και ε, οι ίδιες οι υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες ε, ε, θα αναδιοργανώσουν τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται. Πριν από μερικές ημέρες ανοίξαμε ένα πόρταλ στο οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν πρόσβαση στα μητρώα που φιλοξενεί και νομίζω πως αυτό αποτελεί ένα πρώτο βήμα ούτως ώστε να περάσουμε στην επόμενη φάση όπου θα υπάρχει μεταβίβαση εγγράφων δεδομένων μεταξύ κρατών μελών χωρί αυτό να δημιουργεί περιττέρω άχθο για τι εμπλεκόμενε επιχειρήσει. Και βέβαια όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται με ασφαλή τρόπο, γιατί όταν μιλάμε ε, για δημόσια διοίκηση ή όταν μιλάμε για δημόσιο τομέα υγεία, ε, προφανώ έχουμε να κάνουμε πολύ σημαντικού ε, τομεί οι οποίοι θα πρέπει να παραμείνουν προστατευμένοι. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο, η Αγγέλη Κατομβίνα, έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Να σας συγχαρώ καταρχήν ε, ε, εγώ ε, κυρία Γκάμπριελ, και να σα ρωτήσω. Έγιναν μία σειρά από προτάσει ε, από την πλευρά της Επιτροπής ό,τι αφορά τον ψηφιακό ε, τομέα από την Επιτροπή, αλλά ήταν αλληλεπικαλεπτόμενε αυτέ οι ε, προτάσει. και βέβαια επειδή έχουμε και συναρμόδιε διάφορε επιτροπέ από την πλευρά του Κοινοβουλίου, τελικά ορισμένα αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα, αντιφατικά. Οπότε, τι θα κάνετε σε ό,τι αφορά τι online πλατφόρμες προκειμένου να αποφευθούν τέτοιου είδου αντιφατικέ νομοθεσίε. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Γκάμπριελ έχει το λόγο. Δεν θέλω να μιλήσω εγώ για το πώς θα δουλεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σέβομαι τον τρόπο που το κάνετε έτσι κι αλλιώς. Απλώς από πλευρά της Επιτροπής λέμε πώς καλύτερος συντονισμός μπορεί να επιφέρει και καλύτερα αποτελέσματα. Και αυτό είναι που εξετάζουμε τον πρόεδρο Γιούγκερ με μια πολιτική επιτροπή ακριβώς εφαρμόζοντας αυτό που λέμε ομάδες προγραμμάτων. Με αυτόν τον τρόπο κινητοποιούνται περισσότεροι επιτροποί για περισσότερα χαρτοφυλάκια και όντως στην ανακοίνωση για τις πλατφόρμες κινητοποιήθηκαν οι μισοί επιτροποί. Σήμερα πρέπει να υπάρξει διάρθρωση σε κάθε διάλογο. Και είναι κάτι που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ε, κώδικας διοντολογίας, όλα όσα έχουν να κάνουν ε, με την καταπολέμηση των πλαστών ε, προϊόντων, προστασία των ανηλίκων ε, online. Όλα αυτά τα φόρουμ ακολουθούν διαφορετικές διαδικασίες και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν κοινοποίησεις. Δεν υπάρχει αναρμόνιση. Είναι σε διαφορετική μορφή, οπότε σήμερα αυτό το οποίο λείπει είναι να υπάρχει πιο διαρθρωμένος διάλογος για να μπορούμε να εντοπίσουμε κατευθυντήριες γραμμές. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε νομοθεσία. Το είπαμε, θέλουμε να σεβαστούμε την ε, πολυμορφία, αλλά δεν θα ήταν προτιμότερο να υπάρχει διάρθρωση σε όλους αυτούς τους διαλόγους που στο κάτω-κάτω έχουν κοινό στόχο, την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, προστασία των ανηλίκων. Θα έπρεπε να έχουμε κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες να εφαρμόζονται σε όλες αυτές τις πλατφόρμες και να επιτρέπουν και με μέτρα εθελοντικά αλλά και αυτορύθμισης να επιτρέψουν παραπάνω πρόοδο. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ για συμπληρωματική κύριε Μίνα. Ευχαριστώ. Αναφερθήκατε στο διάλογο και θέλω να σας ρωτήσω τι προσέγγιση θα ακολουθήσατε εσείς στη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους για την σωστή ισορροπία ανάμεσα στις απόψεις τους και τον ε, προβληματισμό που περιλαμβάνεται στην πρόταση. Ευχαριστούμε. Κυρία Γκάμπριελ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έτσι μπορώ να κάνω τη σύνδεση με αυτά που είπα για την προηγούμενη ερώτηση. Θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ την κοινοβουλευτική μου εμπειρία. Πλήρης διαφάνεια στις συναντήσεις με όλους τους αδιαφερόμενους. Δεν υπάρχουν μεγάλοι και μικροί. Δεν υπάρχουν σημαντικοί και λιγότερο σημαντικοί. Μόνο έτσι θα φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου θα φανεί η δυνατότητα, έχοντας ακούσει τα διαφερόμενα μέρη, να πάρω και απόφαση που θα μας βοηθήσει να πάμε προς την κατεύθυνση που και να εντοπίσαμε. Είναι ο πιο απλό τρόπος, με διαφάνεια. Με συνάντηση με όλους τους ενδιαφερόμενους. Να μην δημιουργείται διαχωρισμός. Να μην ξεχνάμε τους στόχους μας και την αντικειμενικότητά μας για να παίρνουμε τις αποφάσεις μας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας. Αυτό ακριβώς θα κάνω. Τίποτα παραπάνω. Ευχαριστούμε. Άξελ Φως για την επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Οριστήσα Επίτροπε, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενισχύσει τη θέση του κλάδου δημιουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αντιμετωπιστεί κυρίως η σημερινή η ανισορροπία ε, που έχει να κάνει με την αξία της δημιουργίας και πώς θα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άνοδο των λεγόμενων fake news, των ψεύτικων ειδήσεων που κυκλοφορούν. Ευχαριστούμε. Απάντηση από την ε, κυρία Γκάμπριλ. Σας ευχαριστώ κύριε Φώσου. Θα επικεντρωθώ στην ερώτησή σας για τη δημοσιογραφία ποιότητας και την καταπολέμηση των fake news, δεν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε πολύ. Δίνω μεγάλη σημασία σε αυτήν τη δημοσιογραφία ποιότητα, γιατί πλουραλιστικά και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης αποτελούν και την εγγύηση για τη δημοκρατία μας. Γιατί μόνο έτσι ο δημοκρατικός διάλογος μπορεί να λάβει χώρα και οι πολίτες, γνωρίζοντας περί τίνος πρόκειται, σχηματίζουν άποψη. Γι' αυτό είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κοινοβούλιο για την πρωτοβουλία αυτή για τις ειδήσει για όλους. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Επιμένω ότι πρέπει να υπάρξει διαπαιδαγώγηση όσον αφορά την δεσογραφία. Πρέπει να επιμείνουμε στις πλατφόρμες και στις επιχειρήσεις ώστε να προωθούν και εκείνες τα μέσα εκείνα που θα μας επιτρέψουν να φτάσουμε σε ειδήσει ποιότητα. για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις δημοκρατικές μας αξίες. Δίνω μεγάλη σημασία και επιμένω σε αυτό. Γιατί έχει να κάνει και με τη θεματική των fake news. Πρέπει να το ομολογήσουμε, δεν είναι νέο φαινόμενο, πάντα υπήρχε. Αυτό το οποίο όμως έχει αλλάξει είναι η ταχύτητα με την οποία διαδίδεται η πληροφορία και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζει τον δημοκρατικό διάλογο και τις αξίες μας. Είναι σημαντικό λοιπόν σήμερα αφενός να διασφαλιστεί ο συντονισμός μέσα από νομοθετικά κείμενα, να δούμε πάλι την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες, για την καταπολέμηση του περιεχομένου του πορνογραφικού ή παιδραστικού, ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αλλά συγχρόνως όλα αυτά τα φόρουμ, τα οποία σας απαρίθμησα, προστασία των ε, ανηλίκων, ε, καταπολέμηση παράνομου περιεχομένου κλπ. Πρέπει να συνδέονται με συντονισμό για να είμαστε αποτελεσματικοί. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να συζητήσουμε καλύτερα και για τη δημιουργία και προστασία δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε κυρία ε, Γκάμπριελ. Συμπληρωματική ερώτηση, όχι, ο κύριος Φως. Ωραία. Επόμενη ερώτηση τότε από τον Νίκολα Ντάντι. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Συγχαρητήρια, Επιτροπέ. Είναι καλό που έρχεται η Επιτροπός. Ελπίζω να μην μας ξεχάσει όταν αναλάβει καθήκοντα. Θα ήθελα να πω ότι εμείς είμαστε ΙΜΚΟ, είμαστε φιλοξενούμενοι και απόψε δεν έχουμε πολύ χρόνο να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Όμως αναφερθήκατε σε πολλά θέματα. Καταρχάς, οι προκλήσεις της ψηφιοποίησης για την αγορά εργασίας. Εμείς ξέρουμε τι ευκαιρίες παρέχονται, αλλά ταυτόχρονα και τι κίνδυνοι υπάρχουν. Εσείς αναφερθήκατε σε πολλά σωστά ζητήματα και δώσατε νομίζω αρκετές σωστές απαντήσεις εδώ στην ακρόαση. Να ρωτήσω όμως ποιες συγκεκριμένε στρατηγικές και δράσεις έχετε κατά νου σε σχέση με τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας το προτάσεών σας για την ψηφιοποίηση και σε ποια φάση βρισκόμαστε. Μετά, για την φορητότητα. Θα ήταν καλό να ασχοληθεί και η Κομισιόν με αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκάμπριελ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντάντη. Και ευχαριστώ που μου δίνετε την δυνατότητα να επανέλθω σε ένα θέμα που θεωρώ πολύ σημαντικό. Πώς συνοδεύουμε την ε, αλλαγή σε αυτό το ψηφιακό κόσμο. Πρώτον, θα συνεργαστώ στενά με την Επίτροπο Τάισεν. Πρώτα απ' όλα για τον κοινωνικό πυλώνα. Η πρόταση υπάρχει ήδη από αυτό το μήνα. Πρέπει να αποφελθούμε από αυτή την ευκαιρία. Δεύτερον, για μένα είναι πολύ σημαντικό σήμερα οι ψηφιακές αρμοδιότητες να μην είναι ψηφιακές αρμοδιότητες βάσεις, αλλά να δουλέψουμε και για τις ψηφιακές δυνατότητες που επιτρέπουν στον άνθρωπο να διακρίνεται από το μηχάνημα. Σίγουρα θα υπάρξουν ε, δουλειές που θα χαθούν ε, γιατί θα τις αναλάβουν τα μηχανήματα. Όμως, ένα μηχάνημα δεν θα μπορέσει ποτέ να δημιουργήσει, δεν θα μπορέσει ποτέ να έχει κοινωνικές σχέσεις. Άρα σε αυτό πρέπει να επενδύσουμε. Γι' αυτό σήμερα χρειάζομαι συγκεκριμένα παραδείγματα από τις χώρες μέλη. Μια πρωτοβουλία που θα στηρίξω είναι ο εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών από το Κοινωνικό Ταμείο. Πρέπει σε κάθε χώρα μέλος να έχουμε ε, τέτοια καλά παραδείγματα και να υπάρχει και συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάτι άλλο είναι το σχέδιο αυτό για τις ψηφιακές δυνατότητες, κατάρτιση για τους φοιτητές. Πρέπει να μπορούν να περάσουν από αυτή την κατάρτιση. Και εδώ θέλω να αναφερθώ και σε κάτι άλλο ευαίσθητο και σημαντικό που έχει να κάνει με τους ανθρώπους που ζουν στην Ήπεθρο. Γιατί θέλουμε να εποφεληθούμε και από τις δυνατότητες των γυναικών για τις γυναίκες συγκεκριμένα τον Οκτώβριο έχουμε την πέμπτη έκδοση του Κότου για το ρόλο των γυναικών στα ψηφιακά. Είναι μια ευκαιρία για να δούμε πως αυτή η κατηγορία πολιτών μπορεί να επωφεληθεί και εκείνη και να βοηθήσει την κοινωνία με τις δυνατότητες που διαθέτει. Ευχαριστούμε κύριε Γκάμπριελ. Α, ναι. Έχετε συμπληρωματική ερώτηση. Παρακαλώ κύριε Ντάντη. Ναι, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα γιατί είδαμε τις επιπτώσεις στην Ευρώπη από καταστάσεις που ζήσαμε πρόσφατα. Θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις. Εμείς είχαμε μια αντίστοιχη οδηγία πάνω στην οποία δουλέψαμε, για την οποία όμως φαίνεται ότι δεν αρκούν αυτά που κάναμε. Έχετε κάτι να αντιπροτείνετε. Ευχαριστούμε κυρία Γκάμπριλ. Δεν ξεχνάω την οδηγία. Είναι το πρώτο νομοθετικό, νομοθετικό μας εργαλείο για την ασφάλεια στον χώρο. Μια από τις πιο σημαντικές πτυχές είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ χωρών μελών. Για μένα αυτό όμως που επίσης είναι σημαντικό είναι ότι με την αναθεώρηση της στρατηγικής θα υπογραμμίσουμε την ανανέωση της εντολής της ΕΝΗΣΑ πώς η υπηρεσία αυτή μπορεί να αποκτήσει πιο σημαντικό ρόλο για την ευαισθητοποίηση ως γραμματεία και ως κέντρο συντονισμού. Περιλαμβάνεται στην σχετική οδηγία. Και κάτι άλλο σημαντικό για μένα, 20 δευτερόλεπτα έχω για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν είναι φυσιολογικό όλα τα εθνικά κέντρα να μην είναι ανοιχτά 24 ώρες, 24, 24 και 7 μέρες τη βδομάδα Αυτά δηλαδή που ασχολούνται με περιπτώσεις ε, κρίσης. Θα έπρεπε. Σε συνεργασία θα έπρεπε να μπορούμε να διασφαλίσουμε τη λειτουργία τους. Χρειάζεται και ένα πρόγραμμα δράσης σε περίπτωση κρίσης. Και αυτό προβλέπεται για το Σεπτέμβριο, ώστε όλοι οι παραγόντες να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν αν υπήρχε κάποιο τέτοιο επεισόδιο. Ευχαριστούμε. Και ερχόμαστε τώρα στην ερώτηση της κυρίας Ρομπέρτα Μετσόλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να μην ε, κάνω δεύτερη ερώτηση, γιατί ίσως έτσι μπορεί να απαντήσει περισσότερο η κυρία Γκάμπριλ. Αυτό λοιπόν που θέλω να ρωτήσω είναι κάτι που απασχολεί πολύ και τους συναδέλφους, είναι η πρόταση για την ηλεκτρονική προστασία. Θέλω περισσότερα να μάθω για την αναγκαιότητα έγκρισης ενός τέτοιου μέσου, μάλιστα αφού έχουμε συζητήσει και έχουμε εγκρίνει τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων. Πού θα συνεχίσετε λοιπόν να διασφαλίζετε με το εργαλείο αυτό την προστασία δεδομένων όταν θα κυκλοφορούν ελεύθερα πια τα δεδομένα. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, η κυρία Κάμπριελ για την απάντηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μέτσολα. Για μένα ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι ότι ακόμα και στην ψηφιακή οικονομία και ψηφιακή κοινωνία είναι λοιπόν να συνεχίσω να υποστηρίζω τις αρχές που υποστήριζα πάντα τα 8 χρόνια που ήμουν μέλος στην Επιτροπή Ελευθερών του Πολίτη εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνω μεγάλη σημασία στις ελευθερίες μας και στα δικαιώματά μας. Πρόκειται για συνέπεια. Ναι, έχουμε το GDPR για του χρόνου και πρόκειται για τα προσωπικά μας δεδομένα. Το e-privacy έχει να κάνει με την εμπιστευτικότητα της διαδικασίας στις επικοινωνίες. Σήμερα είναι εξίσου σημαντικό να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα και για τα άτομα και κατά συνέπεια και την προστασία τους. Το κεντρικό στοιχείο εδώ, και το έχω πει, είναι ο ορισμός της συνένεσης. Η συνένεση του ατόμου είναι και το νήμα που μας καθοδηγεί εδώ. Ο χρήστης δηλαδή πρέπει να δίνει τη συνένεσή του. Αυτό σημαίνει επίσης ότι έχουμε προκλήσεις μπροστά μας. Είναι πολύ σημαντική η συνέπεια, είναι αναγκαία, ώστε οι εθνικές αρχές οι οποίες κοιτούν κατά πόσο τηρείται το GDPR, να μην απομακρυνθούν από το έργο άλλων αρχών που θα φροντίσουν για την τήρηση του e-privacy. δεν πρέπει να υπάρχει επικάλυψη στους στόχους μας. Μη χάνουμε δηλαδή ενέργεια με επικάλυψη. Cookies, πρέβαση by default, αυτά είναι ζωτικά στοιχεία. Και όπως το έχω πει, στο κέντρο βρίσκεται η επιλογή του ατόμου και στη συνέχεια η εμπιστευτικότητα των διαδικασιών. Γιατί θέλω να υπάρχει συνέπεια, υποστηρίζω το εργαλείο αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά κυρία Γκάμπριελ, οπότε έχουμε φτάσει στο τέλος του τμήματος ερωτήσεων και απαντήσεις, απαντήσεων της σημερινής ακρόασης. Ευχαριστώ όλα τα μέλη για τα ερωτήματα που έθεσαν και προφανώς ευχαριστώ θερμά και την ε, κυρία Γκάμπριελ για τα, τις απαντήσεις που μας έδωσαν. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να σας καλέσω να κάνετε μια ε, καταληκτική δήλωση από την πλευρά σας, ε, κυρία Γκάμπρελ, ε, όχι για περισσότερο από πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι. Ο χρόνος περνάει γρήγορα όταν ε, κάνουμε τέτοιες συζητήσεις καθώς όλες οι ερωτήσεις και όλες οι απαντήσεις που δίνονται αφορούν ουσιαστικά ε, ένα κυρίω ζήτημα, το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα την ενιαία ψηφιακή αγορά έτσι ώστε οι κοινωνίες μας, οι καταναλωτές μας, οι επιχειρήσεις μας να μπορέσουν να αναλάβουν εδώ έναν ηγετικό ρόλο. Ε, σήμερα προσπάθησα να σκιαγραφίσω τις κύριες προτεραιότητες από τη δική μου πλευρά και αυτέ είναι καταρχήν ότι θέλω σε κάθε περίπτωση να συμμορφωθώ και να ακολουθήσω τι προτεραιότητε του Προέδρου Γιούγκερ. Από εκεί και μετά, ε, δεύτερη προτεραιότητα είναι η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Η ε, τρίτη προτεραιότητα, να προσπαθώ να βρω συμβιβασμού, να ακούω ε, του ανθρώπου με του οποίου συνδιαλάσσομαι και τους, όλους τους φορείς με τους οποίους συνδιαλασσόμαστε ε, η εμπειρία μου και η μέθοδος εργασίας μου βασίζεται ακριβώς στο διάλογο και τη συνεργασία. Έχω δηλαδή αυτή την ικανότητα του να αφουγκράζομαι τους άλλους. Και άκουσα πολύ προσεκτικά τα όσα μου είπατε εδώ, ε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, και όπως ε, ανέφερα και αρχικά, Είμαι σε κάθε περίπτωση διατεθειμένη να συνεχίσουμε το διάλογο μεταξύ μας. Προφανώς δεν θα ξεχάσω ότι ήμουν, υπήρξα ε, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα, ε, θα προσπαθήσω μάλιστα να δείξω ότι ε, η εμπειρία που αποκόμισα από αυτό εδώ το Κοινοβούλιο που είναι ένα εργαστήριο ιδεών θα αξιοποιηθεί για το καλό των πολιτών μας, για το καλό της κοινωνίας μας. Και έχουμε μία σειρά αποζητήματα να αντιμετωπίσουμε. Ε, και μου μένουν μόνο δύο χρόνια στη θητεία μου. Ε, υπάρχουν ε, νομικές πράξεις που ήδη έχουν υιοθετηθεί και τώρα θα πρέπει να ξεκινήσει εφαρμογή τους μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Θα ήθελα να είχα τη δυνατότητα να σας μιλήσω για την πρωτοβουλία Wi-Fi for Europe, γιατί πραγματικά αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί ένα παράδειγμα απτών ωφελών για τους πολίτες μας. Επίσης, ε, θα ήθελα να είχα περισσότερο, περισσότερο χρόνο να σας μιλήσω για τα δικαιώματα των γυναικών, την κυβερνή ασφάλεια, ε, ε, τις προηγμένες τεχνολογίες, την τεχνολογία των υπερυπολογιστών, των supercomputers, η οποία θα επιτρέψει στην Ευρώπη να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο σε αυτό το τομέα. Ήδη έχουμε επιτύχει σημαντικά επιτεύγματα και έχουμε πολύ δυναμικό ακόμα. Η σημερινή μας ε, συζήτηση καταδεικνύει ε, τις ιδέες ε, που έχουμε και την σαφή εικόνα που έχουμε σε ό,τι αφορά τις αδυναμίες μας, σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και σε ό,τι αφορά τα λία που έχουμε στη διάθεσή μας. Πόσος δρόμος έχει περάσει από την ακρόαση του αδερφού Λικάνεν και τόσες πολλές ερωτήσεις είχαμε τότε στην ακρόαση του που αφορούσαν την ενιαία αγορά, ενιαία ψηφιακή αγορά. Πάντως τα ξανακούσαμε πάλι όλα σήμερα. Είχαμε και την παρουσία πέντε επιτροπών. Αυτό αποδεικνύει πόσο, πόσος χρόνος έχει περάσει σε σχέση με το παρελθόν και πόσο έχουμε προχωρήσει. Γιατί σήμερα έχουμε τα πολιτικά μέσα, τα δημοσιονομικά μέσα, τα διοικητικά μέσα, αλλά κυρίως έχουμε και μία ποικιλία ιδεών και απόψεων που θα μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε τα κοινά ενδιαφέροντα. Και θεωρώ ότι χάρη σε όλα αυτά θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Σήμερα θα πρέπει να κινηθούμε επειδή υπάρχει μεγάλη προσδοκία για αυτό το θέμα στην Ευρώπη. Η ασφάλεια, η αυξανόμενη ισχύ των πλατφορμών, η οικονομία των δεδομένων. Υπάρχουν λοιπόν ξεκάθαρες προτεραιότητες και βλέπω ότι όλες αυτές οι προβληματικές αναφέρθηκαν σήμερα στη συζήτηση. Οπότε ευχαριστώ και πάλι που μου τα υποβάλατε όλα αυτά και μου καταδείξατε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε ακριβώς στο δρόμο που χάραξε ο πρόεδρος Γιούνκερ και να έχουμε μια διαγώνια προσέγγιση. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση ώστε ο συντονισμός και ο διάλογος να δίνουν απαντήσεις πολυδιάστατες, πολυτομεακές, αλλά έχοντας κατά νου πάντοτε το συμφέρον των πολιτών. Επιτρέψτε μου να καταλήξω με κάτι το προσωπικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους γενικούς διευθυντές όλων των γενικών διευθύνσεων και όσους συνέβαλαν στην προετοιμασία της σημερινής μου ακρόασης. Θα ήθελα επίσης να απευθυνθώ σε μια σχολή πληροφορική στο Χάσκοβο, στη Βουλγαρία, που την υποστηρίζω εδώ και 6 χρόνια. Αυτή η σχολή πληροφορική στο Χάσκοβο. Η ψηφιακή τεχνολογία και τα ψηφιακά γραφικά θέλω ακριβώς να βρουν το δρόμο τους στην κοινωνία μας χάρη σε αυτά τα παιδιά και του δασκάλους τους. Ένας παραπάνω λόγος λοιπόν ε, για να μας ε, κάνει υπερήφανους όλους και η Ευρώπη και η Βουλγαρία θα πρέπει υπερήφανη γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Uh, thank you. Thank you very much once again. Σας ευχαριστώ πολύ για μία ακόμα φορά, κυρία Χριστίσα ε, Επίτροπε, για όλε τι απαντήσει που δώσατε, όλα τα σχόλια που κάνατε και για τι δύο ομιλίε σα. Ε, κατά την έναρξη τη ακρόαση και τώρα ε, την καταληκτική παρέμβαση. Ευχαριστώ ε, συναδέλφου συναδέλφους και από τι δύο επιτροπέ και από την Ήτρε και από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδεία, αλλά και από ε, συμμετέχουσε επιτροπέ, ΕΜΚΟ, Γιούρι και ΛΥΜΠΕ. και βέβαια επειδή είχαμε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των δύο διαφορετικών γραμματιών, μπορέσαμε να διοργανώσουμε πολύ αποτελεσματικά τη σημερινή μας ε, συνεδρίαση και θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω και την ε, συνάδελφο Πέτρα Κάμιμπερτε που συμπροέτρεψε εδώ μαζί μου στη σημερινή ακρόαση. Πήγε πολύ καλά, είχαμε πολύ ακριβείς χρόνους ομιλίας και πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που τέθηκαν, και απαντήσεις βέβαια. Το οποίο βέβαια εξαρτήθηκε από τους συντονιστές και των δύο επιτροπών. Σας ευχαριστώ και πάλι θερμά. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ε, και εγώ θα συμφωνήσω πλήρω με τα όσα είπε ο αγαπητό συναδελφό Αιτήριο ε, Μπούζεκ. Δηλαδή, διευκολύνεται πραγματικά τι εργασίε όλων μα ε, εδώ, γιατί όλοι τελικά τήρησαν το χρονοδιάγραμμα τη σημερινή ακρόαση και του ευχαριστώ όλου γι' αυτό. Ευχαριστώ θερμά και την κυρία Γκάμπριελ, η οποία ε, μίλησε για ε, τόσες ώρες σήμερα εδώ. Ευχαριστώ ε, και ε, τις γραμματείες των πύργων Ήτρε και Κούλτ και βέβαια δεν θα ήθελα να ξεχάσω και εκείνου οι οποίοι πραγματικά είναι απολύτως απαραίτητοι χωρίς τους οποίους θα ήταν πολύ δύσκολη η δουλειά μας εδώ στο Κοινοβούλιο, δηλαδή οι διερμηνείς μα, οι οποίοι μετέφρασαν σήμερα το απόγευμα για μα εδώ Τώρα, όπω γνωρίζετε, η ακρόαση αυτή τώρα θα πρέπει να αξιολογηθεί από την πλευρά μα και αυτή η αξιολόγηση θα λάβει η χώρα αύριο ε, το πρωί εδώ, δηλαδή συντονιστέ ε, στι 2 ε, η ώρα στις, των Επιτροπών Ήτρε και Κούλτ θα συζητήσουν το ζήτημα και θα ήθελα να υπενθυμίσω στις συνδεδεμένες επιτροπέ. επιτροπές να μας αποστείλουν τις ε, τοποθετήσεις στο αύριο το πρωί το αργότερο στις 10. Και αν είναι ακόμα στην αίθουσα συντονιστές της Επιτροπής ε, Κούλτ, ε, να τους ζητήσουν να παραμένουν στην για να διευκρινίσουμε κάποια ζητήματα ακόμα. Να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά την οριστή Επίτροπο και σας εύχομαι σε όλους καλό απόγευμα.